Okay, so good afternoon everybody. I hope that you had a nice lunch and I wish... Καλησπέρα σας. Ελπίζω ότι χαρήκατε το γεύμα σας και καλωσορίζω και του αναφέροντες στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Να αναφερθώ λίγο στα όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί συνεδρίασης των ιστών, να σας πω ποιες είναι οι αποφάσεις. Λοιπόν, εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη του Ιουνίου, του Ιουλίου διορθώνει η Πρόεδρος γιατί είμαστε ήδη στον Ιούνιο. Και επίσης ε, συζητήσαμε και για την ημερήσια διάταξη Σεπτεμβρίου, το Οκτωβρίου και το καθεξής. The, the July agenda, namely 0947, 00 οι ε, διερμηνείς σας ενημερώνουν ότι βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω της εργασιακή ε, διένεξη ε, με τη δίκηση για τις συνθήκες εργασίας μας. Καθότι η δίκηση δεν έχει έρθει σε καμία επαφή μαζί μα για την επίλυση τη εργασιακή διένεξη, σα πληροφορούμε ότι η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώ την προβλεπόμενη ώρα λήξη της συνεδρίασης. Προβλέπεται εδώ πέρα η επίγουσα διαδικασία για την 0419. και πήγουσα διαδικασία προβλέπεται μάλλον δεν προβλέπεται και τη 0317. Όσον αφορά τις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις, δεν πρόκειται να συντάξουμε γνωμοδότηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, που είναι έκθεση της Επιτροπής Προπολογισμών, ούτε επίσης για το πρόγραμμα δικαιωμάτων και αξιών, ούτε για την έκθεση ΑΦΚΟ όσον αφορά τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, οι συντονιστές συμφώνησαν να δώσουν στους πράσινους την γνωμοδότηση όσον αφορά τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, εφόσον αποφασίσουν αύριο βέβαια οι βουλευτές της Επιτροπής ΑΦΚΟ ότι θα συντάξουν επ' αυτού έκθεση. Επίσης, ε, εγκρίναμε όλες τις συστάσεις τις οποίες είχα εγώ προτείνει όσον αφορά τις αμφισβητούμενες συστάσεις. Αποφασίσαμε να κλείσουμε κάποιες ε, αναφορές, καθώς επίσης και την 229 θα την κρατήσουμε ανοιχτή. Όσον αφορά τις ρευνητικές επισκέψεις, αποφασίσαμε για τη σύνδεση, σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Άννα το Σεπτέμβριο με έξι μέλη, επικεφαλής αντιπροσωπεία αυτή θα είναι ο Πάλ Ξακή που είναι ο αντιπρόεδρός μας από το ΕΛΚΑ. Τώρα όσον αφορά την... <clears throat> Μάλλον θα αποφασίσουμε τον Ιούλιο για την ακριβή σύνθεση της αντιπροσωπείας αυτής και οι συντονιστές δεν τροποποίησαν τις κατευθυντήρες γραμμές όσον αφορά τις δρευνητικές αποστολές. Αυτό το κάνει η επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Επίσης, αποφασίσαμε να εγκρίνουμε ένα προφορικό ερώτημα και ψήφισμα όσον αφορά τη γερμανική υπηρεσία μέρημνας παιδών Jugendamt και είπαμε να μην ανοίξουμε την αφορά 0775 και 0702 και αποφασίστηκε όλες οι ανοιχτές αναφορές για τα φυτοφάρμακα να προωθηθούν προς την Επιτροπή ΠΕΣΤ προκειμένου να τις επεξεργαστεί ακόμα περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά την ε, συνδιάσκεψη των Επιτροπών Αναφορών ε, στην Γερμανία, αποφασίσαμε εκεί να μην στείλουμε στη διάσκεψη αυτή κάποιον δικό μας βουλευτή. Και επίσης οι συντονιστές ε, λάβανε γνώση των όλων υπόλοιπων σημείων προς ενημέρωση που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Και κατά αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και η συνεδρία των συντονιστών. Τώρα στο σημείο 19 της ημερήσιας διάταξης έχουμε την αφορά 98 για τη στήριξη των ατόμων που φροντίζουν ανάπηρα μέλη της οικογένειάς τους στην Ιταλία. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευθύ αμέσω με την αφορά αυτήν, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τον κύριο Τσίριο, ο οποίος μας είπε τελικά ότι θα ήταν παρόν, αλλά μάλλον δεν θα περιμένω. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στην Μαρία Σιμώνα Μπελίνη. Έχετε το λόγο, κυρία Μπελίνη, για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, την προσοχή που εξακολουθείτε να δίνετε σε αυτή την αναφορά ως Επιτροπή Αναφορών, να σας πω πώς έχει η κατάσταση, τι έχει συμβεί το τελευταίο έτος από τότε που ειδωθήκαμε για τελευταία φορά. Πρέπει παρόλα αυτά να διευκρινίσω ότι το αίτημά μας, η αναφορά μας αυτή, προκειμένου να υπάρχει πραγματικά στήριξη για τα άτομα που φροντίζουν ανάπηρα μέλη της οικογένειάς τους, ισχύει εδώ και 25 χρόνια. 25 χρόνια περιμένουμε μία απάντηση από, την, από τις ταλικές Αρχές. Και το ζήτημα αυτό δεν θα είχε τεθεί ποτέ επισήμω αν η δική σα Επιτροπή Αναφορών δεν είχε επιληφθεί του θέματο, δεν είχε ασχοληθεί με τα όσα έχουν συμβεί στην Ιταλία. Νομίζω πραγματικά θα πρέπει να λάβουμε γνώση του γεγονότος ότι μολονότι δεν μας αφουκράζονται όπως θα έπρεπε στην Ιταλία. Εμείς παραμένουμε, οι φροντιστές δηλαδή, τα άτομα τα οποία έχουν, ε, αν θέλετε, το πιο υποβαθμισμένο επίπεδο ζωής στον δυτικό κόσμο. Και μολονότι στην Ιταλία θα μπορούσαμε να είχαμε άλλες επιλογές για μια πιο αξιοπρεπή ζωή για τα εξαρτώμενα από εμά μέλη, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι καταπατώνται δικά μας και δικά τους θεμελιώδη δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της φροντίδας των εξαρτημένων αυτών ατόμων 24 ώρες το 24ωρο χωρίς να έχουμε άδεια, χωρίς να έχουμε διακοπές, χωρίς να σταματάμε ποτέ. Αυτό το οποίο ζητάμε λοιπόν δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό. Ένα σεβασμό πραγματικά των ανθρωπίνων δικών μα δικαιωμάτων. Αναφερόμαστε στο δικαίωμα στην εργασία, στην ξεκούραση, στι κοινωνικέ σχέσει, στο να μπορούμε να έχουμε επίση πρόσβαση στην υγεία, στην υγειονομική περίθαλψη. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι εμεί φροντίζουμε τα ανάπηρα μέλη τη οικογένειά μα, αλλά δεν μπορούμε να φροντίσουμε εμά του ίδιου, τη δική μα την υγεία. Η κατάσταση λοιπόν αυτή απαράδεκτη υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία, αλλά δυστυχώ όλε οι διατοχικέ κυβερνήσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ουδέποτε διόρθωσαν την κατάσταση και ουδέποτε έλαβαν πραγματικά αποφάσει που θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τα πράγματα και μέχρι σήμερα ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλέ κυβερνήσει που έχουν χρησιμοποιήσει το άλοθη τη έλλειψη δημοσίων πόρων. Χρησιμοποιούν το άλοθη αυτό για να μα πούν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και δεν επιλύουν το πρόβλημα. Θεωρώ ότι οι δαπάνε που θα χρειαζόταν να αναλάβουν οι διαδοχικές αυτές κυβερνήσεις είναι ελάχιστε σε σχέση με το όφελος και το κέρδος που θα είχαμε σε επίπεδο καλύτερη και πιο αξιοπρεπού ζωή για του φροντιστέ. Θεωρώ ότι η φυστάμενη κατάσταση, το να μην προασπίζονται δηλαδή τα δικαιώματά μα, κοστίζει πολύ περισσότερο στο Ιταλικό κράτο από ότι να ίσχυε ένα σύστημα το οποίο θα προέβλεπε μια κάλυψη πραγματικά των αναγκών μα. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, πολλές κυβερνήσεις οι οποίες προσπάθησαν να νομοθετήσουν σε εθνικό, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και παρόλα αυτά βρισκόμαστε αν θέλετε, ως τελευταία χώρα στην όλη αυτή η ιστορία. Γιατί ουσιαστικά είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν προβλέπουν συγκεκριμένε διατάξεις πλαισίωσης και προστασίας των, των ατόμων που αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τα ανάπηρα μέλη τη οικογένειά του. Δεν προασπίζονται, όπω σα είπα, οι νόμοι τη Ιταλία, τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματά μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, να έχουμε πλέον συγκεκριμένες διατάξεις στην Ιταλική νομοθεσία που να μην αποτελούν πλέον απλώς προεκλογικές υποσχέσεις, αλλά να αποτελούν πραγματικές νομοθετικές πράξεις που θα προστατεύουν τους φροντιστές και ιδίω τα πιο ευάλωτα τμήματα του Ιταλικού πληθυσμού. Όταν συναντηθήκαμε σε προηγούμενε συνεδριάσεις θυμάστε ότι είχε προκαλέσει σε πάρα πολλού ε, έκπληξη το γεγονός ότι δεν υπήρχε στην Ιταλία κανένα μέσο στήριξης από το κράτος για τους φροντιστέ, για τα άτομα που φροντίζουν ανάπηρα μέλη τη οικογένειά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ασκηθεί περαιτέρω ποιηση στη νέα πλέον Ιταλική κυβέρνηση προκειμένου επιτέλους να προφηθεί η αναγνώριση της ελάχιστης αυτής προστασίας για τους οικογενειακούς φροντιστές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε συστήματα υποστήριξης, συστήματα κοινωνικών παρεχών και συστήματα υγειονομικής περιθαλψής. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να υποστηρίξουμε τα άτομα αυτά τα οποία λαμβάνουν την πλήρη ευθύνη τη φροντίδα των εξαρτωμένων μελών τη οικογένειά του. Λέμε λοιπόν ω εδώ και μη παρέκει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθούν ιταλικέ νομοθεσίε, οι οποίε θα πλαισιώνουν όχι μόνο τα άτομα αναπηρία, αλλά και του ανθρώπου που τα φροντίζουν. Α μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων να αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστή ειδική κατηγορία στα πλαίσια του Ιταλικού πληθυσμού. Ο Ιταλικό νόμο υπαριθμών 104 που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά ω άλοθη από τι αρμόδιε Ιταλικέ αρχέ, δεν είναι πραγματικό νόμος υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών. Είναι ένα νόμο που έχει να κάνει με την υποστήριξη των ανθρώπων με αναπηρία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εμεί ζητάμε κάτι επιπλέον. Θέλουμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορούμε να ακούμε ως δικαιολογία, ως επιχείρημα ότι έχουμε τον νόμο 104 ή άλλους νόμους. Οι νόμοι αυτοί στηρίζουν τα άτομα αναπηρίες. Αλλά εμείς θέλουμε τώρα ένα νόμο που πραγματικά να πλαισιώνει και να υποστηρίζει του οικογενειακού φροντιστέ, τα άτομα αυτά τα οποία έχουν αναλάβει τη φροντίδα των ανάπηρων μελών τη οικογένειά του. Θα πρέπει και αυτά τα άτομα να πλαισιώσουμε και αυτά τα άτομα να τα φροντίσουμε. Αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να ισχύει σε ένα πολιτισμένο κράτο. Και έχουμε βέβαια και μία καινοτομία τώρα θα λέγω εδώ πέρα, ένα νέο στοιχείο και ολοκληρώνω. Στα τέλη του 2017 καταφέραμε να πετύχουμε τη νομική αναγνώριση σε έναν Ιταλικό νόμο για τους οικογενειακούς φροντιστές. Προβλέπεται επίσης και ένα συγκεκριμένος προπολογισμό, αλλά από την άλλη δεν γνωρίζουμε ακριβώ πώ θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά, τα εθνικά κονδύλια δηλαδή, προκειμένου να στηριχθούν περισσότερο οι οικογενειακοί φροντιστέ. Δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμα 10, 20, 30, ακόμα και 40 χρόνια προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρω αυτή η νομοθεσία αν υπάρχουν κονδύλια τα οποία μπορούν πραγματικά να ε, διοχετευτούν του οικογενειακού φραντιστές αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα από το κράτο μέσω των ε, κρατικών υπηρεσιών και να μην περάσουμε από τρίτου. Θα πρέπει επιτέλους λοιπόν να κλείσει το ζήτημα αυτό και ελπίζουμε ότι με τη νέα κυβέρνηση πλέον της Ιταλίας θα έχουμε μια ειλικρινή πλέον ανταπόκριση στην ανάγκη αυτή που έχουμε εκφράσει τόσο πολλές φορές για υποστήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένατε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ε, για να ακούσετε απάντηση ε, σε, ε, σε όλους τους ισχυρισμούς σας, οι οποίοι είναι απολύτως δικαιολογημένες. Ήλπιζα να δούμε από κοινού τα 19 και 20 σε μια ημερήσης διάταξη και μετά να ακούσουμε τους προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε λοιπόν ε, στην αναφορά 1147 κάθετος 2006 που αφορά περίπου τα ίδια πράγματα, δηλαδή υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικέ παροχέ στα εξαρτώμενα άτομα, άτομα πάσχοντα, ηλικιωμένα, με μαθησιακέ δυσκολίε αυτισμό κλπ. Άτομα που χρήζουν προστασία και φροντίδα δηλαδή. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον, αλλά θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Τσίριο. Σα δίνω το λόγο για 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως, μου ζητήθηκε να εκπροσωπήσω τους αναφέροντες. Πρόκειται για μια αναφορά που έχει να κάνει βέβαια με τα όσα ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά απορρέει από ένα ίδρυμα το οποίο βρίσκεται στο Τωρίνο, που είναι και η εκλογική μου περιφέρεια. Και ουσιαστικά, ήθελα ουσιαστικά να σας παρουσιάσω την αφορά αυτή, γιατί αναφέρον, οι αναφέροντες δεν μπορούν να είναι παρόντες. Πρόεδρε, παρουσιάσατε πάρα πολύ καλά το όλο ζήτημα. Έχουμε εδώ πέρα ένα ζήτημα παρεμφερές με την προηγούμενη αναφορά και νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ένα στοιχειώδη στοιχείο, μια στοιχειώδη πτυχή της αναφοράς αυτής. Καταρχάς, ζητάτε μέσω αυτής της αναφοράς τα εξαρτώμενα άτομα, τα οποία ισχύουν, για παράδειγμα, τα οποία υποφέρουν από μακροχρόνιες ασθένειες, οι οποίοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες που πάσχουν από Αλτσχάιμερ ή από άλλες εκφυλιστικές ασθένειες. Θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να έχουν μια οικονομική στήριξη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας Ιταλίας. Αυτό δεν ισχύει στην Ιταλία ούτε σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί ξέρετε ότι ε, η υγεία στην Ιταλία την χάνει διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο, που μένω από τη μία περιοχή στην άλλη μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η αναγνώριση όμω λοιπόν αυτή, οικονομική στήριξη δηλαδή, που θα έπρεπε να αποτελεί ε, δικαίωμα των ανθρώπων αυτών, δεν καλύπτεται, δεν ε, προασπίζεται ως δικαίωμα στην Ιταλία. Αυτό φάνηκε και από την προηγούμενη αναφορά. Και μέσω της αναφοράς αυτής τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες, μια συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία η γενικότερη δύσκολη οικονομική κατάσταση του ότι έχουν γίνει περικοπές στον δημόσιο προπολογισμό της χώρας. Πέρα από το δίκαιο αυτό, θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το δικαίωμα της οικονομικής υποστήριξης και τα μέλη της οικογένειας του ασθενούς. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν τους ασθενείς διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πολύ συχνά αναφερόμαστε σε αυτούς ως άτυπους φροντιστές. Πρόκειται πάντως για μια παροχή φροντίδα σε οικογενειακό επίπεδο η οποία είναι τεράστια αξίας γιατί συμβάλλει πάρα πολύ στην πιο αξιοπρεπή ζωή του ασθενούς ένας ασθενής, ένα εξαρτόπαινο ουσιαστικά μέλος, ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από μια χρόνια ασθένεια, προφανώς έχει ανάγκη από μια πλαισίωση, από ανθρώπους που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πλαισίωση αυτή, η φροντίδα αυτή, να είναι σύγχρονη και αποτελεσματική. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλουμε να μπορεί να μείνει κατοίκον ο ασθενή και να τον φροντίζει η οικογένειά του. Για να γίνει όμω αυτό, θα πρέπει να καταφέρουμε να στηρίξουμε οικονομικά και να αναγνωρίσουμε όχι μόνο από ηθικής και διοντολογικής πλευράς, αλλά να γνωρίσουμε και στην πράξη τον ρόλο που διαδραματίζουν αυτοί οι οικογενειακοί φροντιστές. Ο ρόλος τους είναι καθοριστική σημασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί, οι φροντιστές, να μπορούν παράλληλα με τη φροντίδα αυτή που παρέχουν στο εξαρτώμενο μέλος να ζουν και τη δική τους ζωή, να έχουν πρόσβαση σε εργασία. Ξέρετε ότι το φαινόμενο αυτό έχει διευθετηθεί σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι στην Ιταλία. Συμφωνώ και εγώ ότι η νέα αυτή κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν σε αυτή, είναι παρόλα αυτά μια νέα κυβέρνηση. Θέλουμε λοιπόν να ελπίζουμε ότι θα κάνουν αυτό που άλλες κυβερνήσεις δεν κάνουν στο παρελθόν. Και όντω ισχύει επιτέλους μια Ιταλική νομοθεσία που αναγνωρίζει τα άτομα αυτά και δίνει επίσης και μια οικονομική στήριξη στους ανθρώπους που φροντίζουν τα εξαρτώμενα μέλη και τους ασθενείς, αλλά δυστυχώς, μόλον ότι έχουμε την νομοθεσία αυτή, λείπουν όλα τα εκτελεστικά διατάγματα, όλες οι άλλες εκτελεστικές νομοθεσίες. Και ξέρετε ότι από τον Ιανουάριο του 2017 υπάρχει μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που κάνει πλέον μία αναφορά στους άτυπους φροντιστές, στην άτυπη αυτή παροχή φροντίδας. Δεν καλύπτονται δηλαδή μόνο η επίσημη φροντίδα η οποία δίδεται από τους νοσηλευτές και τους επαγγελματίε υγείας, αλλά και άτυπη αυτή φροντίδα την οποία παρέχουν οι φροντιστέ σε οικογενειακό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εμπνευστούμε από τις βέρσει πρακτικέ άλλων χωρών σε διεθνέ επίπεδο και να καταφέρουμε τελικά να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό και σε εθνικό επίπεδο στην Ιταλία. Να δώσουμε την προσωπική αυτή αναγνώριση, την ηθική αναγνώριση, αλλά και την επαγγελματική εν τέλει αναγνώριση των ανθρώπων αυτών οι οποίοι θυσιάζουν πραγματικά τη ζωή του για να βοηθήσουν τα εξαρτώμενα μέλη τη οικογένεια του. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσίριο. Να δώσω τώρα το λόγο στην, στον, στην εκπρόσωπο της, Ευρωπα... της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ρίξον Άιτε. Μπορείτε να απαντήσετε και στις δύο ε, αναφορές ε, και στην 98 και στην 1147. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα ε, σε όλους τους αναφέροντες και στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Θα ήθελα να ξεκινήσω επενθυμίζοντας ότι η οργάνωση των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και υγειονομικής περίθαλψης ε, είναι εκτός του τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθείας. Είναι ευθύνη των κρατών μελών και τούτου λεχθέντος καταλαβαίνουμε το ζήτημα της σημασίας των ανθρώπων αυτών που ε, φροντίζουν ε, ε, τα άτομα που, χρειάζονται φροντίδα είναι το δικαίωμα που έχει ο κάθε πολίτης στην μακροχρόνια περίθαλψη καλής ποιότητας. Τώρα αυτό έχει εγγραφεί πλέον στον κοινωνικό πυλώνα ο οποίος προκηρύχθηκε πέρσι, ενώ μεταξύ, μετά ε, την ε, καταχώρηση της, ε, των συγκεκριμένων αναφορών, είναι κάτι στον οποίο, έχουν, το οποίο έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ε, ε, εναρμονίσει, δεν μπορεί να επιβάλλει ε, κανονισμού στον τομέα αυτό, στα κρατη αλλά μέσω της κοινωνικής μεθόδου συντονισμού προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη όταν έχουν θέσει κάποιο σχετικό στόχο προσπαθώντας να επιτύχουν αυτό που είπατε, το δικαίωμα στην μακροχρόνια φροντίδα που θα είναι καλής ποιότητας και προσπαθούμε να οργανώσουμε συνεδριάσεις ομοτύπων, ομοτύπων τα κράτη-μέλη έτσι μπορούν να μάθουν το ένα από το άλλο για τις καλές πρακτικές, μπορούν να δουν το ένα τις καλές πρακτικές του άλλου. Υπάρχουν πολλές μελέτες που μας βοηθούν να εντρυφήσουμε σε διάφορους τομείς για το πώς μπορούμε να παρέχουμε καλύτερη ε, φροντίδα. Ε, συνεργαζόμαστε ε, τώρα ε, και με τον Όσα για να αναπτύξουμε μία νέα μεθοδολογία που θα εξετάζει το πώς μπορούμε να ε, συνυπολογίσουμε το κόστος της μακροχρόνιας φροντίδας και μάλιστα με έναν τρόπο που να επιτρέπει συγκρίσεις. Τα κράτη-μέλη έλαβαν ε, ειδικέ αναχώρασει τάση από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον τομέα τη μακροχρόνια περίθελψη δεν υπήρξαν και πάρα πολλέ συστάσει τα τελευταία χρόνια. Και ο λόγο είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Γιατί για να υπάρξει μία σύσταση πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών δεδομένα και προσπαθούμε τώρα να αναπτύξουμε αυτή τη βάση για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά και να μπορούμε να, επισημάνουμε, να τα επισημάνουμε αλλά μόνο να συντονίσουμε μπορούμε τις προσπάθειες. Εμείς, όπως είπα προηγουμένως, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε καμία πολύ αυστηρή δράση. Ε, Επίση, θα ήθελα να πω ότι κατά το τελευταίο έτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες πρωτοβουλίες ε, για την συμφιλίωση επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου ε, και δόθηκε η δυνατότητα αυτοί οι ανεπίσημοι φροντιστές να λάβουν μία άδεια πέντε ημερών ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Το αποτέλεσμα λοιπόν δεν έχει επιτευχθεί ακόμα, αλλά ε, ε, αυτό έχουμε καταφέρει σε αυτό το τομέα πολιτικής. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ήπια μέτρα, ανταλλαγές πρακτικών, ε, αλλά δεν μπορούμε πέρα από αυτά να παρέμβουμε στα, στα κράτη-μέλη για, τα, για τους τομείς αυτούς. Το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά, αλλά ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Ιταλικό κράτος έχει δεσμευτεί και τώρα εκρεμεί ένα νομοσχέδιο ε, που θα απασχολήσει το νέο κοινοβούλιο για τους οικογενειακούς φροντιστές και έχει, έχει υποβληθεί από το γερουσιαστήκαν Γιάννη στη ε, Γερουσία στις 31 Μαρτίου του 2018. Ας ελπίσουμε να υπάρξουν εξελίξεις, προς το παρόν δεν γνωρίζουμε. Έχετε ξανάρθει όμως από το 2015 εδώ στην Επιτροπή μας και το 2017. Και εμείς ε, ήπια εξουσία έχουμε ως Επιτροπή. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα στα κράτη-μέλη αλλά μπορούμε λίγο να τα πιέσουμε. Και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε και να κάνουμε. Και έχουμε την πρόθεση για να τα ξεδιαλύνουμε λίγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίση μια φανταστική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η στρατηγική βεβαίως δεν ε, σημαίνει πάντα νομοθεσία. Και όπως είπε η κυρία Ριξονάιτε, ε, οι βέλτιστες πρακτικές ε, μπορούν να είναι αντικείμενο ανταλλαγή απόψεων και οι ήπιες αυτές ε, εξουσίες που έχουμε δεν θα πρέπει να μας κάνουμε να λησμονούμε ότι θα πρέπει να πιέζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε μαζί σας. Οι ε, συνάδελφοι, παρακαλώ. Η κυρία Εύη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω εκ νέου τους αναφέροντες ε, που ήρθαν εδώ σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών μία ακόμη φορά, όπως μας υπόθηκε. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται εδώ. Πολλές φορές είχαμε τη δυνατότητα να τους ακούσουμε και να εμβαθύνουμε στο ζήτημα αυτό. Αλλά εδώ και 25 χρόνια δίνουν μάχη και οι άνθρωποι αυτοί αλλά και η Επιτροπή μας προκειμένου επισήμως να αναγνωριστούν οι οικογενειακοί φροντιστές. Θα ήθελα πραγματικά σήμερα να σχολιάσω λίγο την αναφορά αυτή, λέγοντας το εξής. Όλα αυτά τα χρόνια και εγώ πρέπει να σας πω ότι τα τέσσερα χρόνια που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκα με το ζήτημα αυτό και είδα ότι επανέρχεται συνεχώς αυτό το ζήτημα χωρίς να προτείνεται μέχρι σήμερα από την Ιταλική κυβέρνηση μία κάποια λύση, μία σοβαρή δέσμευση προκειμένου να έχουμε ελάχιστη προστασία και ελάχιστη αναγνώριση για τους οικογενειακούς φροντιστές. Σίγουρα πολλές συστάσεις γίνονται και μπορούν να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σαφώ είναι πολύ συγκεκριμένε και περιορισμένε αρμοδιότητε τη κοινότητα όσον αφορά τα εθνικά συστήματα υγεία. Πέρα από αυτό όμω έχουμε και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τη σύμβαση αυτή ω σημείο αναφορά. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τα άτομα με αναπηρίε και με σοβαρέ αναπηρίε μπορούν να ζήσουν με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και αν θέλετε ακόμα και πολύ πιο οικονομικά όταν ζουν κατοίκων και έχουν την άτυπη φροντίδα των μελών της οικογένειάς τους. Δυστυχώς όμως στην Ιταλία ζούμε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία απολύτως προστασία, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς αυτό που μπορώ να πω επί του παρόντος είναι ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει σιγά σιγά να εργάζεται η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας η οποία θέσπισε μάλιστα και Υπουργείο για τα άτομα με αναπηρίες και που είπε ξεκάθαρα ότι ε, θα υπάρχει ε, μία σαφής δέσμευση πλέον της Ιταλικής κυβέρνησης προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε όλες τις πτυχές της αναπηρίας και ιδίω στους φροντιστές και δι τους οικογενειακούς φροντιστές. Ε, μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε μια κάποια πιο συγκεκριμένη και χειροπιαστή ανταπόκριση από την Ιταλική κυβέρνηση και ιδίω μέσω της νέας νομοθεσίας του 2017 που ελπίζουμε ότι θα συνοδευτεί πλέον με εφαρμοστικέ διατάξεις προκειμένου να μπορεί να ισχύει στην πράξη και προκειμένου να μπορεί να ελοποιηθεί προ το συμφέρον όλων αυτών των ανθρώπων που περιμένουν μια απάντηση όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ σαφώ θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. Σαφώ δεν μπορούμε να την κλείσουμε τώρα, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτω ή άλλω θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί και στο μέλλον τι αποφάσει που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη για την προστασία των οικογενειακών φροντιστών. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. I don't... Δεν βλέπω άλλο μέλο τη επιτροπή να ζητεί το λόγο αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω και πάλι ότι το νέο Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να ε, εξετάσει αυτό το θέμα και το νέο νομοσχέδιο για τους οικογενειακούς φροντιστές έχει υποβληθεί στη Γερουσία, από το Γερουσιαστή Καντιάνη, το Μάρτιο και τώρα ε, θα πρέπει να ακούσουμε και πάλι τι έχουν να μας πούν οι αναφέροντες. Ακούσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέλφους. Γιατί αυτό το θέμα πραγματικά πιστεύω ότι ε, ε, είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε να βρεθεί λύση. Και πάλι έχετε το λόγο κυρία Μπελίνη για δύο λεπτά. E Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να διευκρινίσω κάτι. Το έκανε και η Ευρωβουλευτή, η κυρία Εύη, σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής σας. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα των οικογενειακών φροντιστών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Δικαίωμα στην υγεία, δικαίωμα στην ανάπαυση, δικαίωμα στην επαγγελματική απασχόληση. Η έλλειψη πρόσβαση στα δικαιώματα αυτά είναι που δημιουργεί αυτό το υψηλότερο επίπεδο άγχου και την οδύνη ουσιαστικά την οποία βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Όντω εμπιστευόμαστε την νέα αυτή κυβέρνηση, πιστεύουμε ότι θα καταφέρει να επιφέρει μια λύση αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα επαναπαυτούμε. Επίση, ο γερουσιαστή Καντιάνη παρουσίασε ένα νομοσχέδιο όντω, αλλά δεν είναι διαθέσιμο το κείμενο. Επομένω, δεν γνωρίζουμε καν, δυσγνωρίζει γνωρίζει τι εμπεριέχει το κείμενο αυτό, διότι δεν έχει δημοσιευτεί. Αν τελικά εγκριθεί και γίνει νόμος αυτό το νομοσχέδιο, τότε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε πραγματικά να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς. Αυτά τα 60 εκατομμύρια πραγματικά δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουν κανέναν αν ο νόμος αυτός δεν συνοδευτεί από τις απαραίτητες εφαρμοστικές διατάξεις. Και θέλουμε ουσιαστικά να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες ανέφερα. Πραγματική οικονομική υποστήριξη, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ε, και το καθεξής. Θέλουμε να δοθούν συγκεκριμένες χειροπιαστέ απαντήσεις και να μην αποτελέσουν όλα αυτά μία επίφαση, όπως πολύ συχνά γινόταν μέχρι σήμερα στην Ιταλία. Ευχαριστώ. We are not looking for policies. We are δεν ψάχνουμε πολιτικές μέτρα θέλουμε που να αλλάξουν την καθημερινότητα για ε, χιλιάδες ανθρώπους ε, στην Ιταλία με αναπηρίες και ε, τα μέλη των οικογενειών τους. Εμείς δεν θέλουμε ένα χαρτί, ένα νόμο, αλλαγή στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτός είναι ο βασικός στόχος όλου αυτού του εγχειρήματος. Ας επανέλθω λοιπόν για να συνοψίσω και για τις δύο αναφορές. Βεβαίως και θα τις κρατήσουμε ανοιχτέ και θα τις χειριστούμε το ίδιο και τις δύο. Προτείνω να στείλουμε επιστολή ε, στον ε, νέο ε, μέλος της κυβέρνησης, το Λορέντσο Φοντάνα, της ΛΕΓΑ που είναι υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι και παλιός ευρωβουλευτής εδώ, συνάδελφος και θα το ρωτήσω προσωπικά τι γίνεται και θα τον καταστήσω προσωπικά υπεύθυνο για να απαντήσει στο κοινοβούλιο μας και στην Επιτροπή αυτή για υπόλογο το πώς θα ε, αντιμετωπίσουν το θέμα και ποια θα είναι η απάντησή του σε σχέση με το νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη Γερουσία. Και θα τονίσω επίσης ότι δεν θέλουμε να μας στείλουν πια ωραία χαρτάκια, αλλά μέτρα συγκεκριμένα και εξελίξεις θετικέ για τα δικαιώματα των ε, φροντιστών των οικογενειών τους. Αυτό μπορώ να κάνω. Επίσης μπορώ να στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και πάλι και εξηγήσατε ότι νομικός πώς δεν δυνάμεθα, αλλά υπάρχει και ήπια δύναμη η πολιτική είναι η σκληρή δύναμη που είναι ο προπολογισμό και η νομοθεσία, αλλά και η ήπια δύναμη που είναι να πιέζει, να ακού, να μοιράζει ευέλικτε πρακτικές, να προτείνει στρατηγικές κτλ. Θα χρησιμοποιήσω και θα αξιοποιήσω τη δικιά μου ήπια δύναμη και να ζητήσω μια πολύ ειλικρινή απάντηση για το πότε να περιμένουμε λύση για την ε, περίπτωσή σας. Αυτό μπορώ να κάνω και στην Ελεονόρα Εύη, πρέπει να πω ότι το κόμμα σου είναι στην κυβέρνηση. Εδώ, ο κύβος ερήφθη. 25 ε, χρόνια εκκρεμεί αυτή η ιστορία. Λύστε το. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα το κάνετε. <laughs> και μίλε γκράτσι. Χίλια ευχαριστώ σε όλους τους αναφέροντες που ήρθανε. Καλή σας επάνωδο στην ωραία σας χώρα. Προσπαθήστε να υποφεληθείτε από την όχι και τόσο ωραία πόλη των Βρυξελών, να περάσετε καλά όσο είστε εδώ και καλό ταξίδι και ασφαλές. Προχωρούμε. Επόμενη αναφορά. 857. Σχετικά με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα στη Ρουμανία. Και καλώ ορίζουν μια παλιά φίλη, τη Ρωμίνα Αφρασάνη. Ε, με αναφέρουσα. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. αποφασίσαμε να δώσουμε αυτή τη μάχη μαζί. Δεν είστε εδώ για πρώτη φορά, έχετε ξανάρθει. Αλλά σας ευχόμαστε. Το καλώ ορίσατε θερμότατα. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Να σας ευχαριστήσω που με ξανακαλέσατε και μου δίνετε την ευκαιρία να εξακολουθώ να αγωνίζομαι για τα άτομα με αναπηρία στη Ρουμανία και αλλού στην Ευρώπη. Άκουσα τι γίνεται στην Ιταλία και βλέπω ότι υπάρχουν πολλά κοινά ε, στις δύο περιπτώσεις των δύο χωρών. Και πραγματικά έχουν πολλές επιτροπές και οι πολίτες προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το χαρτοβασίλειο εκεί και να δουν τι συμβαίνει. Από τον περασμένο Οκτώβριο που είχα έρθει έχει ε, υπάρξει πληθώρα επιστολών και μεγάλη αλληλογραφία ε, Ρουμανικών Αρχών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχω λάβει και εγώ αντίγραφα. Εμφανίζουν μία ανοθρότητα οι Ρουμανικές ε, Αρχές και αυτό είναι πάρα πολύ αποκαρδιωτικό. Είναι πρόβλημα ε, δεν βιάζονται να το λύσουν. 289 ε, λέει ε, αιτήσει έχουν χειριστεί πέρσι για άτομα με μειωμένο κινητικότητα. Το 98% λέει είχαν θετική έκβαση. Έχω εμπειρία από πρώτο χέρι. Προσπάθησα να ταξιδεύσω στη Ρουμανία σε πολλές πόλεις και αλλού. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα, πρωτοφανή που λένε. Θα ήθελα πραγματικά να δω τις αιτήσει αυτές και πώς ε, ε, έχουν φτάσει στο 98% επιτυχή έκβαση και πώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να ταξιδεύσουν. Γιατί φαίνεται πραγματικά πολύ απίστευτο αυτό και για μένα ε, είναι κατασκεύασμα. Για όσους δεν γνωρίζουν τα πράγματα, από το περασμένο Οκτώβριο Έχω συλλέξει κάποιες φωτογραφίες για να σας δείξω πόσο κακή είναι η κατάσταση και πόσο αδιαφορεί η ρουμανική κυβέρνηση. Και αυτό δεν είναι κάτι που έχω κατεβάσει από το μυαλό μου ή που το έχω ζήσει μια φορά. Είναι η καθημερινότητα ε, των ατόμων ε, αναπηρία, ή προβλήματα κινητικότητα στη Ρουμανία. Θα σας δείξω από ένα σιδηροδρομικό σταθμό φωτογραφίες που το 2015 ε, έχει ε, ανακαινιστεί και, έχουν υποτίθεται ολοκληρωθεί τα έργα πριν από τρία χρόνια και με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι προσβάσιμα αυτά για άτομα με κινητική αναπηρία. Φανταστείτε ότι είστε σε ε, ε αναπηρική πολυθρόνα και θέλετε να πάτε ε, ταξίδι κάπου ανά τη Ρουμανία και τι σημαίνει για κάποιον με αναπηρία και προβλήματα κινητικότητας να προσπαθήσει, να προσπαθήσει να το τονίζω, να ε, ταξιδεύσει στη χώρα. Φτάνετε στο κτίριο λοιπόν Find a ramp. και ε, βλέπουμε μία ράμπα και λέμε «Α, ωραία, θα περάσω από τη ράμπα». φτάνουμε στην πόρτα, αλλά ανοίγει μόνο προς τη μία πλευρά και δεν χωράει να περάσει ένα περική πολυθρόνα. Δεν υπάρχει ε, καθόλου εξοπλισμός και καταστάσεις για να περάσει κάποιος ο οποίος θα πρέπει να ε, αγωνιστεί. Οπότε ε, πολλοί άνθρωποι με αναπηρίες θέλουν να είναι ανεξάρτητοι και περηφανεύονται γι' αυτό, αλλά είστε υποχρεωμένος να ζητήσετε βοήθεια. Εκεί δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει βοήθεια, παρά μόνο συνταξιδιώτης αν έχετε και κάποια στιγμή φτάνετε στην πόρτα. Οι πόρτες είναι κλειδωμένες και δεν μπορείτε να περάσετε. Εδώ οι άνθρωποι δεν ζητάνε τίποτα το εξωφρενικό. Θέλουν να μπουν στο σιδηροδρομικό σταθμό. Κάποια στιγμή μπαίνει, σε πάση περιπτώσει. Πας να βγάλεις εισιτήριο. Άλλη μάχη για να δούμε ποιο κάθεται πίσω από, το, ε, από τη θηρίδα. Μιλάμε για πρακτικά ζητήματα, έτσι. Κάποιο που να μπορεί να θέλει να αγοράσει ένα ειστήριο, να μπορεί να έχει μια ανθρώπινη συζήτηση με εκείνο που κάθεται στον Κισέ και πουλάει τα εισιτήρια. Και τι ανακαλύπτεται όταν απευθύνεστε. Ότι πρέπει 10 μέρες πριν να στείλετε επίσημο αίτημα. Και είναι στη διακριτική ευχαίρεια του σταθμάρχη αν θα ταξιδέψεις. Ας πούμε και σε 48 ώρες πριν, όχι, 10 μέρες. Έχω ταξιδέψει πολύ ε, και με ανεξάρτητο, οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι εντάξει κάπως θα προσαρμοστώ και θα ε, θέλω να ταξιδέψω και θα αποφασίσω τελευταία στιγμή να ταξιδέψω. Ξέρετε ότι συνήθως εδώ υπάρχει θέμα προσβασιμότητας και ακόμα και αν δύσκολο ε, λειτουργούν τα πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα στην αποβάθρα. Άλλα προβλήματα για να φτάσει εκεί δύο τεινά. Θα περάσει απέναντι, αλλά πώς να το κάνεις αν είναι περική πολυθρόνα. Είτε θα πάρεις ένα ε, υπόγειο τούνελ που κατεβαίνει ε, ε, σκάλα. υπάρχει μια πολυθρόνα που είναι κάτω στη σκάλα, αλλά για να ανέβει πάνω να τη χρησιμοποιήσεις χρειάζεται βοήθεια ή αναλκυστήρα. Ε, υπάρχει ένας αναλκυστήρα λοιπόν εκεί στην κλίμακα που δεν ξέρει κανεί να το χειρίζεται. ψάχνεται σε όλο το σταθμό, δεν υπάρχει κανείς. Και πραγματικά εγώ έχω εξαντληθεί να σας τα διαβάζω αυτά και ακόμα δεν φτάσαμε στο τρένο. Και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι στη Ρουμανία. Αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία. Ε, υποθετικά σενάρια. Είναι η πραγματική ζωή. Ε, είναι μια εμπειρία που είχα εγώ προσωπικά πολλές φορές στη ζωή μου και πολλοί άλλοι Ρουμάνοι πολίτες και πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες που θέλουν να ταξιδεύουν στη Ρουμανία. Φτάνουμε λοιπόν στο τρένο, το οποίο έχει αυτή τη μορφή. κάθε είσοδος έχει τρία σκαλιά τουλάχιστον. Και τα άτομα με αναπηρία αγωνίζονται να ανέβουν στο τρένο. Εδώ ένα αρτιμελής που περπατάει κανονικά δεν μπορεί να ανέβει καλά-καλά στο τρένο. Και τώρα μας λέει η Ρουμανική κυβέρνηση ότι το 98% των ενδιαφερομένων ταξίδευσαν. Δεν χωράνε τα αναπηρικά καρατσάκια, δεν μπορείς να μπει. Δεν υπάρχουν φυσικά ούτε κουπέ, ούτε καθίσματα που να προσφέρονται. Όλα αυτά που μας απαντούν είναι στη χώρα του φανταστικού. Τι λένε λοιπόν οι Ρουμανικές αρχές, για ποιο λόγο δεν δίνουν ε, τα στοιχειώδη δικαιώματα σε άτομα μια, ε, ε, με αναπηρία να ταξιδεύουν. Πώς ισχυρίζονται ότι από 289 αιτήσει έχουν ικανοποιηθεί το 98% με τέτοιες συνθήκες. Θα πρέπει να τους τραβήξουμε ταυτή. Όπως είπαν και οι Ιταλοί, και είπατε κι εσείς να ξεφύγουμε από αυτό το χαρτοβασίλειο, να δούμε ε, στην πράξη αποδείξεις πού είναι η προσβασιμότητα. Μην τους αφήσετε να γλιτώσουν με τέτοια κατάφορη περιφρόνηση απέναντι στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που θέλουν να ταξιδεύουν. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, αλλά πρέπει να βγάλουμε μια κόκκινη κάρτα ε, προς την κυβέρνηση της Ρουμανίας και όχι σχέδια και χαρτιά και προγράμματα κτλ. Δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μιλιώση είναι εδώ. Δεν ξέρω, ένα δείχνει τον άλλον. Ποιο θέλει να πάρει το λόγο για να μα εξηγήσει την κατάσταση εκπροσωπώντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι, είμαι Πλαθένθια, ανώτερη εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα αναπηρία και ένταξη ε, των ατόμων με αναπηρίε και θα μιλήσω εκ μέρου τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς ε, αυτά που μας είπε η αναφέρουσα δεν είναι καινούρια. Σας πιστεύω. Σας πιστεύω. Έχω προσπαθήσει να ταξιδέψω με πολλούς ανθρώπους με αναπηρία σε διάφορες ε, χώρες και γνωρίζουμε ε, ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Πραγματικά είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην προστασία των ατόμων με αναπηρίες ε, και στη βελτίωση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών που έχουν εγγραφεί στο πλαίσιο της σύμβασης των ατόμων με αναπηρία και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αναπηρία και, πολλά, και πολλών νομοθετικών μέτρων παίρνει χρόνο. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε χρόνο, δηλαδή έχετε κάθε μέρα να αντιμετωπίσετε ε, αυτά τα προβλήματα και πραγματικά ε, νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα που δεν μπορούμε να επιλύσουμε αμέσως ε, το πρόβλημά σας. Πρέπει όμως να ακολουθήσουμε κάποια βήματα. Το πρώτο λοιπόν που θα ήθελα να κάνω είναι να επενθυμίσω ότι αυτό το ζήτημα προκύπτει λόγω των εξαιρέσεων ε, της ενωσιακής νομοθεσίας 1371 ε, ε, κάποιες υποχρεώσεις αρρωγής μπορούν να αρθούν και ο κανονισμός το επιτρέπει αυτό. Ε, από τότε που εισήχθη η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης ε, ή άρσης ε, των υποχρεώσεων αυτών θα εγκριθεί η πρόταση ελπίζουμε όπως προτάθηκε γιατί πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε έτσι να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα αρρωγής τα οποία έχετε να, έχετε να αντιμετωπίσετε. Βέβαια, έχετε ήδη υπερβεί κάποια, ε, ε, προχωρήσει, γιατί υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την νομοθεσία. Υπάρχει το ζήτημα το πρακτικό της προσπασιμότητας των κτηρίων, των τρένων ε, και θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα ως προς αυτό. Πρώτον, ότι Υπάρχουν οι τεχνικές προδιαγραφές της διαλειτουργικότητας ε, που πρέπει να τις εξετάσουμε πολύ εντελεχέστερα για να δούμε αν υπάρχει έλλειψη συμβατο... Ε, συμμόρφωση, συγγνώμη, αν πρέπει να υπάρξει μια ενίσχυση τους. Υπάρχει και ένας διάλογος αυτή τη στιγμή ε, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων για να δούμε όλες αυτές τις διατάξεις μαζί με άτομα, με συλλόγους που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες, να δούμε αν υπάρχουν συγκεκριμένες προποθέσει ή προδιαγραφέ οι οποίε να είναι προβληματικέ και να προσπαθήσουμε να δρομολογήσουμε ε, τα ε, σχετικά μέτρα. Υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Πράξης για την Κινητικότητα που συμπεριλαμβάνει κάποιες προδιαγραφές ε, για τα κτίρια, όταν τα κράτη-μέλη δηλαδή θα αναπτύξουν την κινητικότητα, υπάρχουν κάποιες, για την προσβασιμότητα, συγγνώμη, ε, πρέπει κάποιες προϋποθέσεις να ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, η κάθετη κινητικότητα. Η κάθετη κινητικότητα πρέπει να εξασφαλίζεται. Πρέπει να πω ότι πράγματι είναι νομοθετικές διαδικασίες ε, χρονοβόρες ε, καταλαβαίνω την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε βραχυπρόθεσμα είναι να ακούσουμε τα εμπόδια τα συγκεκριμένα που έχετε, να τα ε, συγκρίνουμε με τα TSIs, να δούμε κατά πόσο όντως έχουν συμπεριληφθεί, ε, αν απλώς παραβιάζονται. Πρέπει να κάνουμε μία ανάλυση της προσβασιμότητας και των εμποδίων στην προσβασιμότητα. Όμως, όσον αφορά τις νομοθετικές διαδικασίες... Α, κάτι ακόμη, ε, λέει ο Μιλήτρια. Ε, το TSA ισχύει για τις μεγάλες ανακαινήσεις, για τα νέα κτίρια ή για τις νέες υποδομές. Πρέπει λοιπόν να δούμε Ποιε είναι οι προποθέσει που θέτει η νομοθεσία και να το έχουμε αυτό ε, υπόψη μας για τις ε, ε, περχόμενες διαδικασίες. Αναφέρθηκατε στα ταμεία της Ένωσης. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερα γι' αυτό, για να ξέρουμε κατά πόσο οι κανονισμοί έχουν ακολουθηθεί σωστά. Μπορούμε και εμείς να ρωτήσουμε τους συναδέλφους μας. Κάποια από τα ε, ταμεία συμπεριλαμβάνουν κάποιες προδιαγραφές για την ε, προσβασιμότητα. Οπότε είναι χρήσιμο να μεταφέρουμε τους, τους ε, υπεύθυνους συναδέλφους τα σχετικά στοιχεία και να έχετε και κατά νου, όπως είπα πολλές φορές, το ξέρω ότι δεν σας λύνουμε το πρόβλημά σας αμέσως, αλλά ε, θα το είδατε και από τον αριθμό των νομοθετικών μέτρων που προτείνουμε. Πρέπει να βρούμε και διαρθρωτικές λύσει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ακόμη και αν παίρνει περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, για ε, την καταπληκτική σας απάντηση. Πάρα πολύ χρήσιμα και ε, επικοδομητικά ήταν αυτά που είπατε. Οι συνάδελφοι, που δεν είναι και πολλοί, παρόντες στην αίθουσα, ε, είναι εδώ η κυρία Κρούπα, μήπως θέλει να πάρει το λόγο. Μάλλον εσείς και εγώ μόνο είμαστε εδώ. Όχι, δεν θέλετε. Καλά. Τότε να δώσω και πάλι το λόγο στη Ρωμίνα. Μικρόφωνο παρακαλούμε. είναι εκπληκτικό να βλέπω ότι υπάρχει υποστήριξη και να ξέρουμε, το, να, να, ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα κονδύλια. Είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμο. Ε, πριν από τρία χρόνια ε, δόθηκαν αυτά τα κονδύλια και το γεγονό ότι δεν υπάρχουν βασικά χαρακτηριστικά προσφασιμότητα είναι πραγματικά σοκαριστικό. Καταλαβαίνω ότι παίρνουν χρόνο όλα αυτά. Η Ρουμανία δεν είναι όμω καινούριο κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. 11 χρόνια συμμετέχουμε. Ε, υπήρξαν πάρα πολλά εκατομμύρια τα οποία έχουν δοθεί δοθεί στη Ρουμανία για το σκοπό αυτό, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Θα ήθελα απλώ να κάνω έκκληση να ε, συλλεγούν περισσότερα στοιχεία και η Ρουμανία τουλάχιστον να λογοδοτήσει για το πού πήγαν όλα αυτά τα ε, κονδύλια. Να δείξουν τουλάχιστον τι έκαναν προκειμένου να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή για του ανθρώπου με αναπηρία, μια πιο εύκολη ζωή και να του ενθαρρύνουν να είναι ανεξάρτητοι, να ταξιδεύουν. Αυτό θα οδηγήσει βέβαια σε πολλή ευημερία. Ε, βλέπουμε σε άλλε πόσο ενσωματωμένα είναι άτομα με αναπηρία και είναι τόσο κρίμα. Είμαστε πραγματικά πολύ ε, δυσαρεστημένοι που ε, δεν ε, υπάρχει καμία βελτίωση, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν στοιχεία ενσωμάτωσης που μόνο να ονειρευτούμε θα μπορούσαμε. Μπορείτε πάντοτε να βασίζεστε στην υποστήριξή μας, γιατί εμείς πάρα πολλές φορές έχουμε συνεργαστεί για ζητήματα κινητικότητας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια στρατηγική για την κινητικότητα η οποία την αναπηρία, για τα προβλήματα αναπηρίας ε, ε, την οποία θέσαμε σε εφαρμογή και νομίζω ότι είναι πολύ παραγωγική η δουλειά μας. Ας ολοκληρώσουμε τώρα το σημείο αυτό της ε, ημερήσια διάταξη. Έχουμε ζητήσει γνωμοδότηση από την Επιτροπή Τραν. Τη λάβαμε η Επιτροπή Μεταφορών αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο για την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Μεταφορών. Οπότε θα είμαστε σε ε, άμεσο διάλογο με τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών και θα ρωτήσουμε ποιο είναι το επόμενο βήμα που προτίθενται να κάνουν. Άλλωστε, θέλουμε να ε, αποστείλουμε και επιστολή στην ρουμανική κυβέρνηση και να ρωτήσουμε αν αν υπάρχουν στοιχεία για την αξιοποίηση των ενωσιακών ε, κονδυλίων, ε, για να ε, δούμε τι γίνεται με αυτή την πραγματικά πολύ απρόσμενη κατάσταση. Και πρέπει επίσης να τους ρωτήσουμε και πολύ να, να μας ενημερώσουν πώς προχωρούν βήμα προς βήμα για το θέμα αυτό. Όντως υπάρχει πρόοδο στην αναθεώρηση του κανονισμού και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται, πρέπει να φαίνεται και στη Ρουμανία. Αυτά μπορώ να κάνω όμως για την ώρα. Επίσης στείλαμε και ε, μία επιστολή σε όλες τις μόνιμες αντιπροσωπείες στις Βρυξέλλες και τους μιλήσαμε για την κινητικότητα, 29 επιστολές έφυγαν από το γραφείο μας. Είναι ένα ζήτημα ε, επί του οποίου πραγματικά συνεχίζουμε την καλή δουλειά και προσπαθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε να τη συνεχίσουμε. Δεν είναι λοιπόν χαμένος ο δικός σας αγώνας, θα το ε, διατηρήσουμε ανοιχτό το ζήτημα αυτό μέχρι να έχουμε μια θετική απάντηση. Δύο ακόμη συνάδελφοι έχουν έρθει και από ό,τι βλέπω συμφωνούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ε, δείξατε ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να συντονιστούμε, να συνεργαστούμε με άλλους ώστε να μην ε, γίνει μόνιμη αυτή η κατάσταση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Καλή επιστροφή στη χώρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι το υπαριθμό 22 αναφορά 0488 για την παροχή υγειονομική περίθαλψη σε ασθενεί που πάσχουν από το σύνδρομο πολλαπλή χημική ευαισθησία και ηλεκτρομαγνητική ευαισθησία. Δεν είναι εδώ αναφέρον, έχει στείλει όμω επιπλέον έγγραφα. Είναι όμω εδώ εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σα δώσω το λόγο. Κυρία Χέραλντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μα δίνετε να παρουσιάσουμε την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νταϊάννα Χέρολτ ονομάζομαι από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕΤ, Τμήμα Δημόσια Υγεία. Η αναφέρουσα πάσχει από το σύνδρομο πολλαπλή χημική ευαισθησία και το σύνδρομο ηλεκτρομαγνητική υπερευαισθησία. Μα λέει επίση ότι στην Ιταλία δεν αναγνωρίζονται τα σύνδρομα αυτά ω ασθένεια και ότι ε, δεν ε, παρέχεται στους ανθρώπους αυτούς επαγγελματική υγειονομική περίθαλψη. Λοιπόν, ποια είναι τώρα η θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Σας πενθυμίσω καταρχάς τη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίω το άρθρο 168 όπου λέγεται ότι η διαμόρφωση της πολιτικής στον τομέα της υγείας και η οργάνωση του τομέα της υγείας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να νομοθετήσει στον τομέα της δημόσιας υγείας και ούτε δύναται να εκδίδει νομοθετικά μέτρα επί του κλάδου αυτού. Ωστόσο όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί το ζήτημα της ευαισθησίας στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και μπορεί να δίνει συμβουλές και συστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έχουμε για παράδειγμα μέσω της σύστασης του Συμβουλίου για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η σύσταση αυτή δίνει κατευθυντήρες γραμμέ στα κράτη-μέλη. Αλλά η σύσταση αυτή προφανώ δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη-μέλη. Στην ίδια πάλι σύσταση του Συμβουλίου ζητείται από τα κράτη-μέλη σε τακτικό επίπεδο να θεωρούν την πολιτική του όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται αυτό μέσω μια επιστημονική επιτροπή. Η τελευταία έκθεση ήταν του 2015 αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιστημονική Επιτροπή, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επί του παρόντο τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγο να αναθεωρηθεί να αναθεωρηθούν τα ανώτατα όρια προβλέπησή σα του Συμβουλίου. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνεί μέσω διαφόρων μελετών το ζήτημα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, καθώ επίση και τι υπερβεστησίε μπορεί να προκύψει από την υπερβολική έκθεση σε αυτά τα πεδία. Συνοψίζοντα, πρέπει να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να νομοθετήσει στον τομέα τη δημόσια υγεία και ότι η ευθύνη για τη διαμόρφωση των υπηρεσιών δημόσια υγεία, αλλά ακόμα και την αναγνώριση των ασθενειών αυτών, αναπόκειται μόνο στα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Και εμεί σα ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρο. Τώρα μπορούν οι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο, Πέτερ ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα κανονικά αυτό είναι θέμα των Ιταλικών αρχών και να στείλουμε επιστολή να τα λάβει υπόψη όλα αυτά. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι, υπάρχουν συστάσεις όμως προς εφαρμογή τα κράτη-μέλη Αυτά θα πρέπει να λυθούν επί τόπου, να στείλουμε μια επιστολή και να κλείσουμε την αναφορά όταν λάβουμε την απάντηση με το καλό. Αυτή είναι η πρότασή μου, γιατί πραγματικά είμαστε αναρμόδιοι. Exactly. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Και ουσιαστικά και εγώ αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε πια αυτή την αναφορά. Σήμερα πρέπει να γίνει αυτό. Αν δεν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις, αυτό θα κάνουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν την αναφορά. Πολύ ωραία. Και έτσι περνάμε στην επόμενη αναφορά, την υπαριθμό 0853. 0853 λοιπόν, του κυρίου Μάθιου Σπίγκλ, εξ ονόματος του Ιδρύματος Free Morgan, σχετικά με εικαζόμενη μη συμμορφούμενη εφαρμογή και παραβίωση του κανονισμού 338-97 του Συμβουλίου. για τα άγρια είδη χλωρίδας και πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ήρθε από πάρα πολύ μακριά ο αναφέρον. Ακούγεται απίστευτο, αλλά δεν μιλάμε για κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Ήρθε από την Καλιφόρνια και τη Νέα Ζηλανδία ειδικά για τη σημερινή συνεδρίαση. Λοιπόν, σα καλωσορίζουμε ολόθερμα στην Επιτροπή μα. Ουδέποτε έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στη δική μου θητεία, ω πρόεδρο τη Επιτροπή αυτή, να έχουμε καλεσμένου από τόσο μακριά. Πραγματικά τι να πω, θαυμάζω την αντοχή σα. Ήρθατε από τόσο μακριά εδώ πέρα. Και θαυμάζω επίση και την προσήλωση που δείχνει και το ζήτημα αυτό. Κύριε Σπίγκελ, λοιπόν, και κύριε, κύριε Φίσελ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά τουλάχιστον 10 λεπτά. Μην σας πω και λίγο παραπάνω, γιατί ούτως άλλως δεν πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Θα ήθελα να συστηθώ εγώ και ο συνάδελφος Μάθιο έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μελετήσει τις ε, φάλαινες και τα δελφίνια. Ε, όπως είπατε έχουμε έρθει από τη Νέα Ζηλανδία, αλλά είμαι και Ολλανδέζα υπηκός. Ε, συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία από το 2010 με το Free Morgan Foundation. Θα σας πω λίγο περισσότερα γι' αυτό, ε, για την ίδια τη Μόρκα και ο Μάθιου, ο οποίος είναι ο νομικός σύμβουλος ε, έχει έρθει από την Καλιφόρνια και είναι μάλιστα και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ε, Free Morgan ελευθερώστε τη Μόργαν. Να σας συστήσω λοιπόν την ίδια τη Μόργαν. Η Μόργαν ε, είναι μία άγρια όρκα που είναι πολύ περίπλοκη η ιστορία της. Ε, τη βρήκαν στις ακτές της Ολλανδίας ε, και την εχμαλώτησαν. Μπορώ να σας μιλώ για ώρες για αυτό το θέμα. Αλλά θα ήθελα για την ώρα να εστιαστώ όχι μόνο στο περίπλοκο της διαδικασίας, αλλά να καταλήξω στον αναφέροντα. Ε, ή λοιπόν, υπήρξαν χώρες εχμαλώτησης ε, και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε σχέση με τη συγκεκριμένη αναφορά προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στη μεταφορά της Μόργαν από την Ολλανδία στην Ισπανία για κάποια, και για την τεκμηρίωση που χρειαζόταν, κάποια συνοδευτικά έγγραφα ή ε, έπρεπε να ακολουθούν κανονισμοί και νομοθεσία, όπως για παράδειγμα η νομοθεσία σάιτες, η Μόργαν και οποιοδήποτε είδος ε, μπορεί να κρατηθεί με σκοπό να αφαιθεί ελεύθερο μετά στη φύση. Ε, η άλλη επιλογή ήταν ε, να υπάρξει επιστημονική έρευνα η οποία θα γίνει σχετικά με το συγκεκριμένο ζώο. Για να μπορέσουμε να τη μεταφέρουμε χρειαζόταν μια, ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό μεταφοράς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος λέει ότι πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη παρακολούθηση των, των εμπορικών δραστηριοτήτων που αφορούν ε, ζώα τα οποία, ε, των οποίων απειλείται ε, η ύπαρξη, που είναι απειλούμενα με εξαφάνιση. Ε, Πρέπει λοιπόν να αποτρέπεται το ξέπλυμα ε, των ε, ζώων αυτών, δηλαδή να μην κρατώνται ε, σε εχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς. 13 χρόνια είναι η Μόργαν σε εχμαλωσία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα πάρα πολύ πολύτιμο ζώο ε, λόγω ε, των ε, γονιδίων της και για να σας πω γιατί χρήματα μιλούμε λένε, λέει ο τομέας ότι από 1 έως 10 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια στοιχίζει η εμπορική εκμετάλλευση αλλά η Μόργαν συγκεκριμένα θα μπορούσε να στοιχίζει δύο φορές Δηλαδή 10 με 20 εκατομμύρια δολάρια είναι ένα από τα πιο πολύτιμα ζώα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο. Ε, για να μπορέσω λοιπόν να σας το θέσω σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό, 10 όρκες υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και η Μόργαν είναι η μόνη η οποία είναι άγρια όρκα. Ε, στην, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει πολύ σοβαρά το λαθρεμπόριο των άγριων ειδών. Ε, υπάρχει ένα σχέδιο δράσης μάλιστα, το οποίο συμπεριλαμβάνει την ιδέα ότι το λαθρεμπόριο αυτό είναι ένα από, τα, ε, πιο, από τις πιο κερδοφόρες εγκληματικές δραστηριότητες παγκοσμίων. Ε, τρεις βασικοί, τρία, τρεις βασικοί άξονες, η μεγαλύτερη επιβολή, η καλύτερη προστασία ε, και η ε, αποτροπή. Ε, όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι περισσότεροι μπορεί να θεωρούμε ότι το λαθρεμπόριο των άγριων ειδών σημαίνει ότι πηγαίνουν και παίρνουν τα ζώα και τα βάζουν μέσα σε μια βαλίτσα και τα μεταφέρουν. Όμως Ουσιαστικά το εμπόριο αυτό μπορεί να σημαίνει ότι για παράδειγμα ε, συμμετέχουν σε διάφορα σόου τα ζώα και κάποιος πουλάει εισιτήρια για αυτά τα σόου. Ε, από τα ζώα που σώζονται, ε, τα άγρια είδη, ε, εχμαλωτίζονται. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία για τα οποία γίνεται αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ε, ζώα τα οποία ε, αφορά όλη αυτή η υπόθεση, παρά το γεγονό ότι αντιμετωπίζουμε, ότι δεχόμαστε το γεγονό ότι δεν έχει να κάνει με την ευημερία η συγκεκριμένη αναφορά, παρόλα αυτά έχουν πολύ σημαντικέ συνέπειε για την υγεία και τη ζωή αυτών των ε, ζώων. Ε, η Μόργαν βλέπετε πόσο έχει πληγώσει μόνη της τον εαυτό τη λόγω του στρε, του άγχου που έχει, γιατί βλέπετε εδώ πούμε την πληγή επειδή χτυπάει στο κλουβί ή ε, ε, έχουν τα ούλα της καταστραφή επειδή μασάει το, το τσιμέντο. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και ο συγκεκριμένος κανονισμός του Συμβουλίου 338 κάθετο 97 που είναι κατά τη αδικαιολόγητης εχμαλωσίας των άγριων ειδών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής που μας δίνετε την ευκαιρία και τον επιπλέον χρόνο. Πραγματικά το εκτιμούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό να ανεβάσω την παρουσίασή μου. So we're here today with three... Έχουμε τρία αιτήματα βασικά σήμερα. Πρώτον, να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Δεύτερον, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει το πιστοποιητικό του σχέδιό του και το θέμα να παραπευθεί στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μια οριστική ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου. Γιατί αυτές οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο τη Μόργαν, αλλά οποιοδήποτε εμπορεύεται αυτά τα είδη. Υπάρχουν ε, προβλήματα στην μεταφορά της νομοθεσίας ε, δηλαδή όλες οι όρκες δεν έχουν δημιουργηθεί ε, ίδιες, ίσες. Υπάρχει ε, το παράρτημα Α και το παράρτημα Β. Το παράρτημα Α αφορά την άγρια όρκα που έχει γεννηθεί στη φύση και το δεύτερο την όρκα που έχει γεννηθεί σε εχμαλωσία. Τα άγρια είδη πανίδα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για πρωτογενώ εμπορικού σκοπού. Ο κανονισμό του Συμβουλίου 338 είναι ένας βασικός κανονισμός που εφαρμόζει τη σύμβαση CITES στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα το άρθρο 8.1 και το 8.3. 8.1. Η ε, επίδειξη στο κοινό για εμπορικούς σκοπούς, για κέρδος κτλ ε, ε, θα απαγορεύονται όσον αφορά το παράρτημα α. Τελεία. Από εκεί ε, απαγορεύεται οποιοδήποτε εμπόριο ειδών ε, στο παράρτημα Α, ακόμα και αν είναι σε εχμαλωσία, είδη που έχουν γεννηθεί άγρια. Το άρθρο 8.3 προβλέπει κάποιες εξαιρέσει. Εξαιρέσει από την απαγόρευση μπορεί, δύνανται να εκχωρηθούν, δεν οφείλουν ε, βάσει ενό πιστοποιητικού και κατά περίπτωση. Είναι πολύ περιοριστικό αυτό και θα πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Άρα λοιπόν βάσει το άρθρο 8, του 338, η εξαίρεση ε αφορά την πρόοδο της επιστήμης, η F ε αφορά τον πολλοπλασιασμό ή την αναπαραγωγή, 8.3G έρευνα ή εκπαίδευση, 8.3G είναι το πιστοποιητικό της Morgan για έρευνα ή ε, εκπαίδευση. Είναι μία σελίδα όλο και όλο το πιστοποιητικό. Είναι πολύ απλωστευτικό το έντυπο. Το 2001 λοιπόν υπήρξε μια γενική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σύμφωνα με την ομολογία του δικαστηρίου οι εξαιρέσεις θα πρέπει να ε, ερμηνεύονται περιοριστικά. Αυτό λέει και το άρθρο 8.3 που προβλέπει ε, απόκληση από τη γενική απαγόρευση πάρα πολύ στενή λοιπόν η ερμηνεία και περιοριστική. 865-2006 λέγεται ο εφαρμοστικός κανονισμός και το παράρτημα 5 έχει αυτό το έντυπο ε, που είναι το πιστοποιητικό για τις εξαιρέσεις και είναι και η άδεια μεταφορά του ε, βάσει του άρθρου 9.2. Και πάλι λοιπόν, τι είναι ειδική η περίπτωση η Μόργαν είναι ένα θηλυκό ζώο που γεννήθηκε στη φύση, εχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε από την Ολλανδία στην Ισπανία με χρήση αυτού του εντύπου. Και το πιστοποιητικό, η εξαίρεση ε, περιγράφεται σε μία γραμμή. 18-8. Και τελικά έχουμε μια περιγραφή συγκεχημένη, ε, κάθετος ε, συμπυκνωμένη, κάθετος ασαφή. Ότι χρησιμοποιείται, λέει, για την πρόοδο της επιστήμης, ε, κάθετος για πολλαπλασιασμό, κάθετος για εκπαίδευση ή έρευνα. Όλα αυτά μαζί το ίδιο πρόβλημα στη μεταφορά της νομοθεσίας ε, διαιωνίστηκε όταν το 2012 αναθεωρήθηκε το έντυπο. Σε μια πρόσφατη απόφαση του αρμόδιου πρωτοδικίου στην Ολλανδία, η ημερομηνία 22 Απριλίου, 26 Απριλίου, ε, λέει το δικαστήριο ότι το πιστοποιητικό της Μόργαν έχει εκδοθεί βάσει το άρθρο 8.3G ε, του βασικού κανονισμού ε, με σκοπούς ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς και καμία άλλη εξαίρεση. Ε, συμπέρασμα και επιπτώσεις τώρα. Θα, θα πρέπει να εξηγούνται για να γίνουν κατανοητές εξαιρέσεις, όχι απλώς να αναφέρονται. Ε, γιατί αυτό οδηγεί σε ε, σύγχυση. Άρα λοιπόν οι, Ολλανδικές αρχές και οι Ισπανικές επικαλούνται μόνο τη γραμμή 18-8 για να δικαιολογήσουν ότι δεν απαγορεύεται η αναπαραγωγή. Ποια αναπαραγωγή, αφού είπαμε ότι χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς. Είπε λοιπόν το Ραδικό Δικαστήριο ότι αυτή η διατύπωση δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις εξαίρεσης. Άρα λοιπόν για τις χειριστικές αρχές του σάιτες, για να μπορέσουν να επιβάλλουν την νομοθεσία θα πρέπει να καταλάβουν τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Αλλά ε, υπάρχει πρόβλημα γιατί στο ποιητικό δεν είναι ξεκάθαρο το τι επιτρέπεται γιατί όλα αυτά είναι ε, στο ίδιο κουτί όπου μπορείς να τσεκάρεις διάφορες επιλογές και αυτό οδηγεί σε σύγχυση. Και το ζώο τώρα ακιοφορεί, η Μόργαν. Ε, το 2015 όταν μεταφέρθηκε δεν ήταν έγκυος. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι. Επειδή είναι του, του παρατήματος Α. Και ζευγάρωσε με ένα είδος αρσενικό, ε, ε, ε, ένα αρσενικό ζώο από το παράρτημα Β που έχει γεννηθεί στην εχμαλωσία. Και τι γίνεται τώρα με το φαλενάκι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και για να αποφευθούν, ε, να αποτραπούν στο μέλλον τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται να επιβληθούν κυρώσεις και μάλιστα ε, υποχρεωτικές. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούν κάποιοι ένα ζώο με και ως ε, δεν επιτρέπεται. Άρα λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, επαναλαμβάνω, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει το σχέδιο του εντύπου πιστοποιητικού και να παραπευθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μια οριστική ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Πρωτού δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή μας δεν έχει αρμοδιότητες ε, προκειμένου να παραπέμψει το ζήτημα αυτό στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δύνατο να το κάνει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν το κρίνει αναγκαίο. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να παραπέμψουμε οποιαδήποτε υπόθεση οπουδήποτε. Δεν είμαστε δικαστική επιτροπή. Δεν έχουμε τέτοια δικαστική αρμοδιότητα. Πάντως χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε ότι έχετε και αυτή την πρόθεση, αυτή την επιθυμία. Σα το λέω εξ αρχή πάντω για να μην απογοητευτείτε με εμά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα το, λίγο, το λόγο έχει ο κύριο Ροντρίγκε Ρομέρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να τονίσω ότι οι διατάξεις στις οποίες αναφερθήκαμε τώρα δεν έχουν να κάνουν με την σύμβαση ΣΑΙΤΕΣ για το Διεθνές Εμπόριο Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας. Δεν έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της σύμβασης αυτής, αλλά ουσιαστικά έχουν να κάνουν με νομοθεσίες και διατάξεις που ισχύουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμαστε δηλαδή για συμμόρφωση ουσιαστικά με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίποτα παραπάνω. Όπως ε, είπαν και αναφέροντες, οι διατάξεις αυτές ισχύουν ήδη από το 2001. Υπό το φως αφορά σε αυτής εξετάσαμε περισσότερο την εφαρμογή των διατάξεων αυτών για τη χρονική αυτή περίοδο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να εντοπίσει στη χρονική αυτή περίοδο κάποια σημαντικά προβλήματα με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Δεν έχουμε εντοπίσει κανένα πρόβλημα στην εκτενέστατη αυτή μελέτη που έγινε το 2007 όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία των ειδών άγρια πανίδα και χλωρίδα για τον έλεγχο του εμπορίου του δηλαδή. Επίση, τα κράτη-μέλη στι τακτικέ εκθέσει που υποβάλλουν ε, όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του κανονισμού δεν έχουν γύρει κανένα τέτοιο ζήτημα στην αυτό το οποίο ανέφεραν οι αναφέροντε και ούτε εν τέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον μέχρι στιγμή, έχει δεχθεί κάποια υπερδοποίηση από κάποιο άλλο συμβαλόμενο μέρο. Για τα ζητήματα αυτά τα οποία θίγουν στην αφορά του οι αναφέροντε. Παρ' αυτά, Υπό το φως αναφοράς αυτής και των όσων ακούσαμε και υπό το φως όλων αυτών των επιχειρημάτων ήρθαμε σε επαφή με τα κράτη-μέλη προκειμένου να έχουμε μία περαιτέρω ανάλυση και παρακολούθηση των όσων ισχύουν σε εθνικό επίπεδο και το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιο διαρθρωτικό πρόβλημα με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων του εφαρμοστικού κανονισμού. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω επίση ότι έχουμε χιλιάδε άδειε σε αιτήσια βάση που εκδίδονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χιλιάδες πιστοποιητικά και άδειε σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό του Συμβουλίου όσον αφορά το διεθνές αυτό εμπόριο. Μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις εφαρμοστικές διατάξεις, όπως μας είπαν οι αναφέροντες, και ότι όντως δεν καταλήγουμε και εμείς, δεν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπονομεύεται η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού μέσω των εφαρμοστικών διατάξεων σε κανένα επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια μεμονωμένε περιπτώσει σαν αυτή που χρησιμοποιήσει ο αναφέρον, προκειμένου να υπογραμμίσει περισσότερο τα επιχείρηματά του, αλλά υπάρχουν ε, εθνικά ένδικα μέσα για να επιληθούν τα ζητήματα αυτά που νομίζω ότι έχει χρησιμοποιήσει ούτω ή άλλω ο αναφέρον στο οικείο κράτο μέλο ή στα οικεία μάλλον κράτη-μέλη. Υπενθυμίζω ότι η αλλω ο αναφερον στο οικειο κρατο μελος η στα Επιτροπή δεν ήθιστε να ασχολείται με μονομένες περιπτώσεις, αλλά επικεντρώνεται περισσότερο σε διαρθρωτικά εμπόδια τα οποία μπορούν να προκύψουν στην εφαρμογή ενός κανονισμού και τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δεν συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης τέτοιων εμποδίων ή τέτοιων αδυναμιών όσον αφορά την εφαρμογή των λόγων καονισμού. Σας ευχαριστώ. Thank you Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Ποιο είναι ο πατέρα του παιδιού, αυτό το μικρό φαλενάκι. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Κοιτάξτε, δύο ε, αρσενικές φάλαινες ενδεχομένως μπορεί να είναι ο πατέρας. Ε, έχουν μια επιθετική στάση. Ε, η μία από αυτές τις φάλαινες επιτέθηκε σε έναν εκπαιδευτή. Ο άλλος πιθανός πατέρας φάλαινος αστικά σκότωσε έναν εκπαιδευτή και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή τέλο πάντων, επειδή ακριβώ ανήκουν, όπω σα είπαμε, σε ξεχωριστή κατηγορία. Α μην το αναλύσουμε περισσότερο το ζήτημα. Ίσως θα πρέπει να μιλήσουν πρώτα ευρωβουλευτέ και θα σα δώσω το λόγο για να δευτερολογήσετε. Η κυρία Στέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εδώ και ο Χαβιέρ Αλμούνια που ζήτησε το λόγο και εκπροσωπεί το Europark, αλλά είναι κυρίως αντιπρόεδρος ε, της ε, αρμόδιας ε, και, ε, Ένωση Ζωολογικών Κήπων στην Ισπανία. Ζήτησε να μιλήσει, αλλά η, η, πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί να μιλήσει. η απάντηση ήρθε τη Δευτέρα και είχε βγάλει τα ειστήρια και έχει έρθει. Είναι αντιπρόεδρο της Ιβυρική Ένωσης Ζωολογικών Κήπων. Αυτό το θέμα έχει φτάσει στην Επιτροπή Αναφορών, είχε ε, ψηφίσει, είχε αποφασίσει. Η Όρκα Μόργαν είναι ένα ζώο που έχω δει στο Europark πριν από τρία χρόνια. Ε, Θα τα θυμάται πολύ καλά ο Πέτερ Γιάρ γιατί το συζητήσαμε πάρα πολύ την περασμένη θητεία και πριν από τρία χρόνια πήγα σε αυτό το πάρκο. Η Ολλανδική κυβέρνηση ζήτησε από την Ισπανική κυβέρνηση να αναλάβει αυτή την όρκα. Υπήρξε δικαστική απόφαση και η Επιτροπή μας θεώρησε ότι όλα ήταν εντάξει, όπως έλεγε και η δικαστική απόφαση. Τώρα επανερχόμαστε με αυτό το θέμα και θέλω να σας πω ότι η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι σωστή και καλωσορίζω και εγώ τους αναφέροντες γιατί η έρευνα σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει έρευνα αναπαραγωγική. Δεν το λέει πουθενά αυτό ο κανονισμός ότι δεν μπορεί να κεωφορήσει το ζώο. Λένε οι αναφερόμενοι ότι λάθος έχει ερμηνεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα παντού σε όλα τα κράτη-μέλη λένε ότι οι σάιτες ερμηνεύεται σωστά και δικαιώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγικούς ερευνητικούς σκοπούς. Και ε, στην Ουτρέχτη ε, όταν εκδικάστηκε η απόφαση, ε, η υπόθεση μάλλον, κατέληξε ε, στην απόφαση το δικαστήριο ότι μπορεί να κυοφορήσει η Όρκα Μόργαν. Το Σεπτέμβριο θα γεννήσει. Ε, δεν ξέρουμε ποιο από τα δύο αρσενικά είναι ο πατέρας. Την ελέγχουν, την παρακολουθούν πάρα πολύ. Αν ήταν στην ανοιχτή θάλασσα θα είχε ε, αποβιώσει και οι σάιτες της Ολλανδίας και οι σάιτες της Ισπανίας συντονίζονται και ερμηνεύεται τώρα με λάθος τρόπο τον κανονισμό. Υπάρχουν δικαστικές αρχές, κυβερνητικές αρχές και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το λέει γι' αυτό. Θα παρακαλούσα να κλείσει αυτό το θέμα. Να χαρούμε για τον τοκετό το Σεπτέμβριο. Είναι και κουφή επίσης. Και επειδή οι, όρκες διαλέγονται, συνομιλούν με τα μέλη της οικογένειάς τους με κάποιο τρόπο, με κάποιους ήχους, ε, η ίδια αυτή η Μόργαν είναι κοφή. Να δούμε πώς θα επικοινωνεί με το φαλενάκι της. Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ ωραίο, ας μην το, ας μην το ασχημένουμε. Ε, υποστηρίζουμε την Ιβηρική Ένωση Ζωολογικών Κήπων και όλων ε, όλους εκείνους που τα υποστηρίζουν όλα αυτά για να πάνε καλά. Και να μην έχουμε παρερμηνίες, γιατί ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε οι αρμόδιες αρχές, ούτε οι σάιτες Ολλανδίας, ούτε οι σάιτες Ισπανίας καταλήγουν εκεί. Και είναι η δεύτερη φορά που το συζητούμε εδώ. Και θέλω να υποστηρίξω απολύτως τον Χαβιέρα Αλμούνια και την σωστή ε, ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν δεν είχε την τύχη αυτή η όρκα Μόργαν, σήμερα δεν θα υπήρχε και θα μιλούσαμε για πολύ χειρότερη έκβαση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστούμε κυρία Εύη, το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ δεν συμφωνώ με τα όσα είπε η συνάδελφος μόλις τώρα. Ουσιαστικά θα ήθελα να στηρίξω τα όσα ζητάνε οι αναφέροντες. Και αυτό διότι πέραν των όσων μας είπανε, το πώς δηλαδή μπορούμε να έχουμε καταλήξει μέσω νομοθετικών κενών ή παράκαμψη της νομοθεσίας σε μια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα άγριο είδος ουσιαστικά, το οποίο μεταφέρθηκε από την Ολλανδία στην Ισπανία. Εκεί δόθηκε ένα πιστοποιητικό και τώρα βρίσκεται σε εκμαλωσία και χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Πραγματικά ενώ, ενώ, ενώ στο πιστοποιητικό λέγεται ότι χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς κτλ. Πραγματικά λοιπόν, δεδομένων όλων αυτών, δεν νομίζω ότι μπορούμε να εθελοτυφλήσουμε. Ας δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Χρησιμοποιείται ένα άγριο είδος το οποίο θα έπρεπε να προστατεύεται και όχι να χρησιμοποιείται για εμπορικού σκοπούς και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι όχι μόνο χρησιμοποιείται, κυοφορεί κιόλα. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει σαφώς να καταφέρουμε να αποτρέψουμε άλλα τέτοια φαινόμενα στο μέλλον, δηλαδή να χρησιμοποιούνται άγρια είδη για κερδοφορία ουσιαστικά, για λόγου οι οποίοι είναι σαφώ κερδοσκοπικοί. Λοιπόν, θα πρέπει όχι μόνο να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, αλλά να διευκρινίσουμε και λίγο περισσότερο αυτό που μα είπαν ή αυτό που μα ζήτησαν οι αναφέροντε. Όλα αυτά τα πιστοποιητικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασαφέστατα και οδηγούν πάρα πολύ συχνά σε παρανοήσει. Εμεί δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωμοδοτήσει, όπω το είπατε και εσεί, κυρία Πρόεδρε, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το κάνει αυτό γιατί πολύ συχνά προσφεύγει ουσιαστικά στο Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου αυτό να αποφανθεί για την ερμηνεία τη κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερη ε, ερμηνεία όσον αφορά τι διατάξει τη ε, κοινοτική αυτή νομοθεσία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γιούζο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι αν αυτή η όρκα δεν είχε μεταφερθεί στο Λόρο Πάρκε, ε, θα είχε πεθάνει γιατί είναι κοφή. Και όπως γνωρίζετε ε, ζουν ε, σε κοπάδια οικογένειες και επικοινωνούν με ήχους. Θα, δεν θα ζούσε, είναι κουφή η όρκα. Και καλά που είναι στο Λοροπάρκε και, και δεν έχει χάσει τη ζωή της κιόλας. Το θέμα αυτό επανέρχεται ξανά και ξανά. Και το κάνει αυτό το Ίδρυμα Free Morgan Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα και το μοναδικό που το επαναλαμβάνει σε 38 σελίδες συνοψίζεται σε μία φράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μεταφέρει σωστά τον κανονισμό 338 το 97 ε, στα αντίστοιχα έντυπα από τους επόμενους κανονισμούς. Και σύμφωνα με αυτό το Ίδρυμα τα συγκεκριμένα έντυπα δεν αντανακλούν σωστά ε, τις απαγορεύσεις των διαφόρων ε, κανονισμών, το 338, το 8 άρθρο κτλ. Αυτή είναι δική τους ερμηνεία, γιατί όλα τα κράτη-μέλη, τα δικαστήρια, τα Ολλανδικά και οι υπόλοιποι τους διαψεύδουν και δεν τους δικαιώνουν. Είναι μια δική τους ερμηνεία και επιμένουν και έρχεται και πανέρχεται γιατί θέλουν να αλλάξουν τον κανονισμό. Δεν έχει νόημα πια αυτό. Θα πρέπει ο κανονισμός να γίνει όπως θέλουν αυτοί. Πουθενά δεν λέει ότι μια όρκα που χρησιμοποιείται για επιστημονικούς σκοπούς δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ε, ε, αφού τους λένε τα δικαστήρια όχι. Τους λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όχι που μόλις την ακούσαμε και τα κράτη-μέλη δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο θα πρέπει εδώ να συζητάμε το ίδιο θέμα και να το γυρνάμε γύρω-γύρω. Ας την κλείσουμε γιατί μετά από δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πρέπει να ξαναπούμε ότι είναι κακοί οι κανονισμοί και πρέπει να το, τους αλλάξουμε όπως αρέσει σε αυτό το Ίδρυμα. Ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε φτάνει πια μέχρι εδώ. Ευχαριστώ. I don't have any more members that... Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να πάρει το λόγο. Οπότε να δώσω και πάλι το λόγο με χαρά στον κύριο ε, Σπίντελ και την ε, ε, δόκτωρα Φίσα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούμε τι, λέτε, τι μας λέτε, με σεβασμό. Δεν συμφωνούμε. Με την εξαίρεση βέβαια της συναδέλφου σας που μας υποστήριξε. Στις 18 ε, Απριλίου υπόθηκε στο δικαστήριο ε, ότι υπήρξε παραβίαση, ε, ότι δηλαδή δύο ξεχωριστά άδρα συνδυάστηκαν σε ένα και υπήρξε ένα πιστοποιητικό το οποίο σκοπό είχε μόνο επιστημονική έρευνα αλλά όχι αναπαραγωγή. Δεν λέω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να κλείσει αυτή η αναφορά λόγω του αιτήματο του Λόρο Πάρκ. Ε, εμείς ε, αφιερώνουμε χιλιάδες ώρες της, από το χρόνο μας. Δεν έχουμε κανένα απολύτως όφελος από το να τελεσφορήσει αυτή η κατάσταση. Είναι όμως κάτι το πολύ θετικό για τα ζώα, όχι μόνο για τη Μόργαν, ε, υπάρχουν χιλιάδες ζώα ε, τα οποία πλήττονται από όλη αυτή την υπόθεση, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή εμείς απλώς έχουμε παρακολουθήσει ένα συγκεκριμένο ζώο από τη στιγμή της εχμαλωσίας του μέχρι σήμερα, μπορούμε να δούμε πού έχουν γίνει τα σφάλματα και ενδεχομένως απλώς δεν τεκμηριώνει κανείς τι συμβαίνει σε πολλά από τα υπόλοιπα ζώα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Εντάξει, είναι κουφή η Μόργαν και θα είχε πεθάνει στην άχρια φύση. Λάθος είναι αυτό. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα μέρη στα οποία θα μπορούσε να είχε πάει η Μόργαν. Εμείς είχαμε προτείνει να πάει αρχικά ε, σε ένα χώρο που θα επιπλέει στον οργανισμό, ε, στον ωκεανό, συγγνώμη. Εκεί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα δελφίνια και πολλές άλλες φάλαινες στην ίδια κατάσταση. Διαφορετικά θα μπορούσε να είχε πάει σε κάποιο είδους καταφύγιο για πολλού λόγους λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το έχουμε συζητήσει αυτό σε πολλά δικαστήρια. Οι αποφάσει είπατε ότι ήταν πάντοτε αντίθετες με εμά. Όχι δεν ισχύει αυτό. Συχνά τα δικαστήρια συμφωνούσαν με την επιχειρηματολογία μας αλλά είπαν στο τέλο ότι δεν θα γινόταν καμία μεταφορά της Μόργαν από εκεί που ε, βρίσκεται. Ε, μόνο το Ολλανδικό δικαστήριο ε, αποφάνθηκε κατά κάποιο τρόπο εναντίον μας. Ο κύριος Σπίγκελ, μας ρωτήσατε ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της Μόργαν. Το θέμα είναι ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ε, του μπαμπά της του μπαμπά του παιδιού της Μόργαν. Ο SeaWorld είναι οργανισμός που είναι ιδιοκτήτη ε, ε, το Δεκέμβριο του 2017 μεταφέρθηκε ε, η Μόργαν, είχε ήδη γίνει σύλληψη, ήταν ήδη έγκυος, ε, και τότε μεταφέρθηκε ο πατέρας. Ε, έχουμε όλα τα έγγραφα. Ε, ο ένας υποψήφιος πατέρας είχε έγγραφα που έρχονταν από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ο Sea World έκανε μία απαγόρευση αναπαραγωγής όταν είπε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες, δεν θα υπάρξει αναπαραγωγή άλλων ορκών και γι' αυτό ακριβώς απαγορεύτηκε ε, η αναπαραγωγή της Μόργαν που βρισκόταν στο Λόρο Πάρκ. Λόρο Πάρκε. Ε, δηλαδή η Λόρο Πάρκε ήξερε ότι υπήρχε μία απόφαση της SeaWorld να σταματήσει η απαγόρευση. Παρόλα αυτά, επειδή πολλούσαν εισιτήρια, συνέχισαν με την διαδικασία ε, της πώλησης εισιτηρίων και μάλιστα επέτρεψαν την αναπαραγωγή της, ε, γνωρίζοντας την απόφαση της SeaWorld. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς ε, να πει ε, ότι σωστά ε, έγινε η εφαρμογή των άρθρων του κανονισμού. Σε διαφορετικές παραγράφους λέγονταν διαφορετικά πράγματα τα οποία απλώς συγχωνεύτηκαν και με όλο το σεβασμό που τρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνετε λάθος, τα στοιχεία που δίνετε δεν είναι τα πραγματικά Όντως υπάρχει ένα, μια σύγκρουση συμφερόντων, γιατί εμείς ε, έχουμε αναφέρει ένα ζήτημα με, με, την εχμαλωσία των ζώων από τότε που ξεκίνησε ε, ο κανονισμός και μετά άρχισε να υπάρχουν, να υπάρχουν, διάφορα προβλήματα ερμηνείας, όχι μόνο της συγκεκριμένη υπόθεσης, αλλά και διαφωνίες σε σχέση με την ερμηνεία του εφαρμοστικού οργανισμού ε, και σε σχέση με τον κανονισμό του Συμβουλίου. Ω πρόεδρο τη Επιτροπής μα τώρα βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι πολύ λίγα τα παρόντα μέλη για να ψηφίσουμε. Χρειάζεται απαρτία 12 μελών για να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Τώρα έχω μέλη που ζητούν να κλείσει αναφορά και άλλα που ζητούν να παραμείνει ανοιχτή και δεν μπορώ να κάνω ψηφοφορία. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι παρόντες βουλευτές. 12 χρειαζόμαστε για απαρτία για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Και αυτή τη στιγμή πώς είμαστε. 7. Και τέρμα. Δεν μπορώ να ψηφίσω αυτή τη στιγμή. Πράγμα που σημαίνει 8. 8. 12 πρέπει να είμαστε για ε, να ψηφίσουμε. Και έχουμε και αποκλίνουσες απόψεις. Και δεν βοηθάει το γεγονός ότι είναι σύσσωμο σχεδόν το ΕΛΚ εδώ, γιατί δεν μπορώ να κάνω ψηφοφορία. Χρειαζόμαστε 12 άτομα. Άρα θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρητά να διερευνήσει το θέμα εάν ε, συνάδει και συμμορφώνεται με τη σύμβαση ΣΑΙΤΕΣ, δηλαδή αν επιτρέπεται να αναπαράγονται ε, οι όρκες εχμαλωσία ε, όταν το ποιητικό τους λέει έρευνα και εκπαίδευση. Και θα επανέλθουμε όταν έχουμε απαρτή, αλλιώς δεν μπορώ να προχωρήσω. and, and that is it. Μίσης Εσταράς. Η κυρία Εσταράς. Κοιτάξτε, να γραφεί στα πρακτικά ότι πάνω από ένα μήνα ξέραμε ότι είναι αυτή η συνεδρίαση σήμερα, όπως και οι αναφέροντες. Η ομάδα μου είναι εδώ και ο Πέτερ Γιάρ συντονιστής. Έχουμε έξι μέλη παρόντα και είναι και ομάδα EFTD, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ε, αφήσει, ε, έχουν παραμελήσει μάλλον τις υποχρεώσεις τους. Εμείς είμαστε εδώ πλειοψηφία, αλλά οι απόντες έπρεπε να είναι παρόντες και να λένε ε, την άποψή τους. Γιατί έχει έρθει ένας κύριος από την Τενερίφη, όπου βρίσκεται το Λόρο Πάρκε. Έχουν έρθει από μακριά οι αναφέροντες ε, και το Λόρο Πάρκε πραγματικά προσέχει και φροντίζει την όρκα, την έγκυο ε, και την ευημερία των ζώων και τα λοιπά και αξίζει καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα η ομάδα μου έχει την πλειοψηφία για να κλείσει αυτό και να μπορέσουν να παρακολουθούν την όρκα με την ησυχία τους ε, ε, στο Λόρο Πάρκε. Εδώ πρόκειται για παραμέληση λοιπόν ευθυνών και η ομάδα μας που έχει την πλειοψηφία δεν μπορεί να κερδίσει γιατί δεν υπάρχει απαρτία. Θα πρέπει να τους ανακαλέσετε στην τάξη. Δεν μπορούν να εγκαταλείπουν έτσι τις ευθύνες τους και κάποιοι να κερδίζουν απόντες και ε, οι παρόντες να χάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Of course we will reflect this in the minutes. This... Ναι, βεβαίως θα το γράψουμε αυτό στα πρακτικά, αλλά μπορώ να σας πω εγώ είμαι η πρόεδρος της Επιτροπής εδώ και τέσσερα χρόνια και ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν έχει συμβεί να μην μπορέσω να ε, κάνω ψηφοφορία λόγω της ε, αμέλεια των υπολείπων ομάδων. Η πράσινη δεν είναι εδώ. Η Γκουε που ζήτησε να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συγκεκριμένη αναφορά δεν είναι εδώ. Και αν δεν υπάρχει απαρκία που να επιτρέπει την ε, ψηφοφορία, τότε παραπέμπεται η απόφαση στους συντονιστές. Αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό πρέπει να κάνουμε βάσει των κανόνων μας. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που βλέπω. Κύριε Μάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση μόνο, διαδικαστική. Ε, ομολογώ άγνοια εδώ. Αν κάποιος ζητάει να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή και η πλειοψηφία ζητάει να κλείσει. Και εφόσον δεν ψηφίσουμε, γιατί υπερισχύει η άποψη να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, ενώ η παρούσα πλειοψηφία ζητεί να κλείσει. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπερισχύει η μειοψηφούσα άποψη. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε για να το καταλάβουμε όλοι, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. It would have been very simple. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ απλό αν είχαμε μία άποψη μόνο, αλλά υπήρξε και μία άλλη άποψη που εκφράστηκε από την κυρία Εύη και είπε ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και άλλη μία από, άποψη που εκφράστηκε από τους συναδέλφους που είπαν ότι θέλουν να κλείσει αυτή η αναφορά. Αυτή, σε αυτή την περίπτωση γίνεται ψηφοφορία και σε αυτή την περίπτωση δεν έχω απαρτία 12 μελών που σημαίνει ότι δεν μπορώ να διεξαγάγω ψηφοφορία. Ε, ε, ακολουθούμε λοιπόν στο το σημείο 15 του κανονισμού που λέει ότι πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτή για την ώρα και να την παραπέμψουμε και πάλι στους συντονιστές για να υπάρξει απόφαση. Πέτερ. Λοιπόν, θα παρακαλέσω και πάλι εσείς ως πρόεδρος να επιπλήξετε ε, τις ε, απούσες πολιτικές ομάδες. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Και μάλιστα όταν κάποιοι ζητούν να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και δεν πατάνε στη συνεδρίαση, ε, αυτό δεν είναι συμπεριφορά. Να το διαβιβάσετε αυτό στις ομάδες που σήμερα λάμπουν δια της απουσίας τους, διότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και είναι και ασέβεια απέναντι στους αναφέροντες. Η δημοκρατία ζει από τη συζήτηση και θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν, κυρίως εκείνοι που ήθελαν να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη αναφορά. Και καταλαβαίνω και τη δική σου οργή, ούτε εσύ είσαι χαρούμενη με τις εξέλιξεις αυτές, σε βλέπω. Είμαι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα τέσσερα χρόνια που προεδρεύω τέτοια κατάσταση να έχω να αντιμετωπίσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προεδρεύσω βάσει των ε, κανόνων ε, του εσωτερικού ε, κανονισμού, δηλαδή λαμβάνουμε την απόφαση παραπομπής στους συντονιστές και θα αποφασιστεί στην ερχόμενή μας συνεδρίαση τον Ιούλιο. Εν τω μεταξύ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε αυτό το πολύ μακρύ ταξίδι. Σας ευχαριστούμε όλους που όλους ενδιαφέρεστε για αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον ενδιαφέρον ζήτημα της Μόργαν. Σας ευχαριστούμε για όσα κάνετε και για όλα όσα δεν έχετε ακόμη κάνει και θα συνεχίσετε να κάνετε. Είτε εδώ είτε αλλού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και καλό ταξίδι. Και πριν πάω στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξη, πρέπει να πω ότι έχουμε το καλύτερο, την καλύτερη δυνατή γραμματεία. Εκπληκτική δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που προετοιμάσατε σε δευτερόλεπτα ε, τη δουλειά μας, ώστε τουλάχιστον να ε, ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό σωστά. Πάμε λοιπόν ε, στην αναφορά 392-2015, ξενόματος οργάνωσης Compassion in World Farming, συμπόνια στην παγκόσμια κτηνοτροφία. Με 18 υπογραφέ οργανώσεων προωθούν την ορθή μεταχείριση των ζώων, την ορθή μεταχείριση των αγελάδων γαλακτοπαραγωγή. Δίνω το λόγο στον αναφέροντα για 5 λεπτά. Να περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να αποχωρήσουν όσοι αποχωρούν. Okay, so Mr. Κύριε Στίβενσον, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Στην έκθεση του Πέρση, ο καθηγητής Μπρουμ είπε ότι οι αγελάδε γαλακτοπαραγωγής και η ευημερία τους ίσως είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό την έννοια αυτή έχω απογοητευτεί για τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απάντησή της προς εσάς στις 28 Μαρτίου που είπε ότι την παρούσα φάση δεν θεωρεί απαραίτητο να αναλάβει οποιαδήποτε περαιτέρω δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πολύ χρήσιμο εργαστήρι τον περασμένο Οκτώβριο για τα κράτη-μέλη. Και αυτό θα πρέπει να ειδωθεί ως εφετηρία για τη δουλειά που χρειάζεται έτσι ε, ώστε να προσαρμοστούμε με την οδηγία 98 58 και όχι το τέλος της προσπάθειας. Um, now, η οδηγία 98-58 ρίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι διοκτήτες ε, κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε τα ζώα τους να ε, ζουν σε ευημερία και να μην προκαλούνται ε, δεινά, βασανιστήρια, πόνος ή τραυματιστή χωρίς λόγο. Το Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια χρήσιμη έκθεση για την ευημερία των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και κατέδειξε κάποια σοβαρά προβλήματα. Είπε ότι τα τελευταία 40 χρόνια η γαλακτοπαραγωγή ανά ε, αγελάδα έχει διπλασιαστεί και παραπάνω και αυτό οδηγεί σε κάποια προβλήματα. Μεταξύ αυτό ε, υπερμεγέθης μαστούς με ειδήματα και πολλές αγελάδες έχουν μεταβολικά νοσήματα. Η μαστίτιδα είναι μια λίμωξη πάρα πολύ επώδυνη του μαστού της Αγελάδας και η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι η μαστίτιδα είναι καθημερινό φαινόμενο στις γαλακτοπαραγές ε, Αγελάδες. Και ε, βεβαίως και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα ε, είναι ο τοκετός. Και πολλές και η χολότητα και πολλές ε, αγελάδες που χωλένουν ε, πονούν πάρα πολύ. Ε, έχουμε λοιπόν πολλά έλκη, πολλούς τραυματισμούς και πολλές φορές τα κλουβιά στα οποία ζουν οι αγελάδες είναι πάρα πολύ στενά ή πάρα πολύ κοντά, βραχαία δηλαδή. Άρα τα πίσω τους πόδια είναι σε διαδρόμους και τραυματίζονται καθώς ε, όταν προσπαθούν να σηκωθούν ή να ξαπλώσουν, ε, προσκρούν στα τυχώματα των κλωβών ή στα κάγκελα. Σε πολλά κράτη-μέλη κρατούνται ε, ενσταυλισμένες οι αγελάδες και δεμένες όλο το χρόνο και 24 ώρες το 24ωρο. Αυτή είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεμβρίου και έχει όλη αυτή, αυτή την ε, ιδηλιακή, βοκολική ε, φωτογραφία. Αλλά πολλές από τις αγελάδες αυτές δεν έχουν δει στη ζωή τους λιβάδι, δεν έχουν βοσκήσει σε εξωτερικό χώρο. Ε, το Νοέμβριο που μας πέρασε κάναμε μια έρευνα σε νέα γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις για την παραγωγή τυριού γκράνα παντάνα. Ε, ήταν σοκαριστική η εικόνα των αγελάδων. Ποτέ δεν βόσκησαν στο εξωτερικό. Ε, ήταν σταυλισμένες ε, και ε, ε, πολύ απεισχνασμένες οι περισσότερες. Ε, όπως σας είπα, η ίδια έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τα δικά μας στοιχεία τι δείχνουν. είμαστε ε, απογοητευμένη από την ε, απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα συμπεράσματά της ότι στην παρούσα φάση δεν θεωρεί σκόπιμο να αναλάβει νέα δράση. Βεβαίως και χρειάζεται δράση. Και καλούμε και επιμένουμε και πιέζουμε την Επιτροπή σας, παρακαλούμε αφήστε ανοιχτή την αναφορά μας και επίσης σας παρακαλούμε, ζητήστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους και τα κράτη-μέλη να δουν ποια βήματα θα πρέπει να αναλάβουν για να συμμορφωθούν με την οδηγία 98 κάθετος 58 που προβλέπει ότι θα πρέπει να αναβάνονται όλα τα μέτρα έτσι ώστε να ε, εξασφαλίζεται η ευημερία των αγελάδων και να μην προκαλούνται άσκοπα τραυματισμοί, βασανιστήρια και πόνος. Επίσης, κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εκδοθούν ε, ή εκδόθηκαν ε, για την κοπή της ουράς των χείρων, των μικρών χειριδίων. Ε, και για τις αγελάδες χρειάζονται να γίνουν κάποια βήματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Στίβενσον. Η κυρία Γκούσμα είναι η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΑ. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Θα μιλήσω πολωνικά. Φορέστε λοιπόν τα ακουστικά σας. Szanowni Państwo, e, zgodnie e, z tym, co powiedział e, Pan... Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσαμε από τον κύριο Στίβενσον, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει σημαντική εργασία για την βελτίωση της ευζοίας των ε, αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όσον αφορά το καθαρά νομοθετικό τμήμα. Εδώ πέρα βασιζόμαστε στην οδηγία 98 58 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ζώων στα εκτροφία. Και αναφερόμαστε επίσης και σε ένα κανονισμό του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004, υπ. 82, όσον αφορά τα επίσημα μέτρα ελέγχου όσον αφορά πάντα την ορθή μεταχείριση των ζώων εκτροφής. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα σαφέ νομοθετικό πλαίσιο, σαφή νομοθετικά μέτρα, τα οποία εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να στηρίξει τα κράτη-μέλη ω προ την εφαρμογή τη ενωσιακή νομοθεσία, αλλά η επιβολή και η εφαρμογή των μέτρων αυτών εμπίπτει πάντα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμεί έχουμε κάνει πολλού ελέγχου πάντω. Ήδη το 2013 κάναμε δύο ελέγχους, δύο επιθεωρήσεις στην Φιλανδία και την Αυστρία. Και εν συνεχεία το 2015 κάναμε πέντε τέτοιες επιθεωρήσεις στον Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, την Εσθονία και στην Αυστρία. Στόχος των επιθεωρήσεων αυτών ήταν να δούμε αν τελικά εφαρμόζεται στην πράξη το νομικό αυτό εργαλείο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν είναι το πλέον ιδανικό και κατάλληλο και αν όντω συμβάλλει στην ορθή μεταχείριση των ζώων και αν όντω αποτρέπει την βάναυση μεταχείρισή τους. Οι εκθέσεις μετά τον έλεγχο, οι οποίες συντάχθηκαν, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει των πέντε αυτό επιθεωρήσεων και ελέγχων έχει συνταχθεί μάλιστα και μία έκθεση αξιολόγησης, η οποία καταλήγει στα εξή συμπεράσματα. Λέγεται στην έκθεση αυτή ότι επί του παρόντος τα κράτη-μέλη έχουν στη διάθεσή τους εύλογα νομικά μέσα προκειμένου να συμβάλλουν στην ευζοία των ζώων εκτροφής. Και μάλιστα προβλέπονται τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά μέσα, καθώς επίσης και κυρώσεις σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και κώδικες δεοντολογίας πάντα σε εθνικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής εν συνεχεία συζητήθηκαν τον Οκτώβριο του 2017 με κάθε δυνατή λεπτομέρεια σε ένα εργαστήριο που έφερε τον τίτλο «Καλύτερη κατάρτιση για πιο ασφαλή τρόφιμα» το οποίο συνοργανώθηκε, μάλλον οργανώθηκε, από την ε, Γενική Διεύθυνση Σάντε και έλαβε χώρα στην Ιρλανδία αυτό το εργαστήριο. Πολλοί εμπειρογνώμονε από διάφορα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν σε αυτό το εργαστήριο και μπόρεσαν κατά αυτόν τον τρόπο να τριφύσουν περισσότερο στα διαθέσιμα ένομα μέσα τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ επίση και σε όλου του δείκτε συγκριτική αξιολόγηση που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτίμηση τη ορθή μεταχείριση των ζώων εκτροφής. Τονίστηκε επίσης επανειλημμένος ότι τα κράτη-μέλη είναι τα πλέον αρμόδια στον τομέα αυτό και ότι έχουν στη διάθεσή τους μια ολόκληρη εργαλειοθήκη που τους επιτρέπει πραγματικά να βελτιώσουν τις συνθήκες μεταχείρισης των γελάδων γαλακτοπαραγωγής. Προφανώς χρειάζονται ακόμα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να εμπλακούν όμως τη δικασία αυτή και οι ίδιοι οι γαλακτοπαραγωγοί, καθότι είναι οι πλέον ενδιαφερόμενοι στην όλη αυτή διαδικασία και αυτή είναι η πλέον υπεύθυνη για την ορθή μεταχείριση των αγελάδων γαλακτοπαραγωγή. Μετά από όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ήδη έχουν συμβεί πολλά σημαντικά όσον αφορά την αναθεώρηση και την αξιολόγηση τη κατάσταση τη ευζοία των αγελάδων γαλακτοπαραγωγή. Επομένω, δεν μπορούμε παρά να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία και να προσθέσω επίσης το σημείο αυτό ότι πέρυσι, τον Ιανουάριο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε μια πλατφόρμα για την ευζοία των ζώων, Animal Welfare Platform, οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα αυτή μάλιστα συνεδρίασαν τον Ιούνιο, αυτό το μήνα δηλαδή, και είχαμε και μάλιστα πολλούς εκπροσώπους από τα κράτη-μέλη που συμμετείχαν στην πλατφόρμα αυτή, αλλά και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ίδιου του παραγωγικού κλάδου. Και θεωρώ ότι μάλλον αυτό είναι το καλύτερο δυνατό φόρουμ που έχουμε αυτή τη στιγμή για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε αυτό το τομέα, της ευζοίας των ζώων δηλαδή. Τώρα υπάρχουν και δύο υποομάδες οι οποίες έχουν θεσπιστεί. Μάλλον μία υποομάδα διορθώνει ο μιλητής, είναι επιχειρησιακή και μάλιστα άρχισε να λειτουργεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και έχει να κάνει με τη μεταφορά και τη μετακίνηση των ζώων. Και έχουμε και μία ακόμα υποομάδα η οποία θα θεσπιστεί σε λίγες μέρες και θα έχει να κάνει με τους χείρους. Πρόκειται για επίσημα λοιπόν πλέον όργανα που θα έχουν ως βασικό ρόλο να συντάξουν τους μελλοντικούς κανονισμούς και τις μελλοντικές κατευθύνσεις γραμμές Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα μας, επιτρέψουμε, θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε την ορθή μεταχείριση των ζώων τώρα. Δεδομένου του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιορισμένες αρμοδιότητες, μάλλον συγγνώμη, έχει περιορισμένους ε, πόρους, και η μονάδα η οποία είναι υπεύθυνη για την ευζοία των ζώων έχει πεπερασμένους πόρους που σας είπα και πολύ μικρό προσωπικό. Θα ενθαρρύναμε τα μέλη της ευρωπαϊκής αυτής πλατφόρμας να θεσπίσουν ε, τις δικές τους ομάδες, όχι επίσημες υποομάδες, αλλά άτυπες αν θέλετε ομάδες που θα μπορούσαν να ασχοληθούν περαιτέρω με το ζήτημα αυτό και να προτείνουν βελτιώσει όσον αφορά την ευζοία άλλων ειδών όπω τα άλογα και η σκύλη. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Αναφερθήκατε σε μια πλατφόρμα. Σε ποια πλατφόρμα αναφέρεστε. Δεν κατάλαβα, λέει η Πρόεδρος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πλατφόρμα. Σε τι ακριβώ αναφέρεστε. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα. Μα αναφέρθηκα στην πλατφόρμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευζοία των ζώων, κυρία Πρόεδρε, η οποία θεσπίστηκε πέρυσι μετά από απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η πλατφόρμα θεσπίστηκε τον Ιούνιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο, λέει τώρα η ομιλήτρια, και μάλλον η πρώτη συνεδρίαση έγινε τον Ιούνιο, η δεύτερη έγινε τον Νοέμβριο και στις 21 Ιουνίου την Πέμπτη θα έχουμε την τρίτη συνεδρίαση της πλατφόρμας αυτής. Ο Επίτροπος Αντριουκαίτης θα είναι παρόν. Βλέπω εδώ επίση και κάποια ενεργά μέλη της πλατφόρμας αυτής, στην συνεδρία της Επιτροπής σας. 75 πάντως είναι οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα αυτή, εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη, αλλά εκπροσωπείται επίσης και ο παραγωγικός κλάδος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς επίσης και ιδιώτες εμπειρογνώμονες. Και επί του παρόντος η πλατφόρμα αυτή, πρώτον, απέδειξε πραγματικά την αξία της, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και όντως προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και προωθεί επίσης κάποιες νέες ιδέες. Ωραία, κατάλαβα τώρα. Πολύ καλά, πολύ καλά έκανα και έθεσα το ερώτημα αυτό, γιατί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μια διακομματική ομάδα όσον αφορά την προστασία των ζώων, στην οποία συμμετέχουν ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες θα μπορούσε και η δική μας η διακομματική ομάδα να συμβάλλει σε αυτή την όλη εργασία. Ας μην μακρηγορήσουμε όμως περαιτέρω. Ας ακούσουμε τώρα τα μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Εύη πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. προκύπτει από όλες αυτές τις έρευνες, τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που γίνανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από διάφορους οργανισμούς αλλά και από ακτιβιστές και έπειτα και από τους επίσημους ελέγχους φαίνεται τελικά ότι η εντατική κτηνοτροφία των αγελάδων γάλακτοπαραγωγής γίνεται σε πολύ δεινές συνθήκες τελικά όπου βλέπουμε ότι έχουμε στάβλους όπου στηβάζονται πάρα πολλές αγελάδες, ότι οι συνθήκες υγιεινής στις μονάδες αυτές εκτροφής είναι άθλιες, δεν τηρούνται τα ελάχιστα πρότυπα και είδαμε και στις φωτογραφίες ότι υπάρχουν πάρα πολλές αγελάδες γαλακτοπαραγωγής οι οποίες ουδέποτε βόσκουν σε βοσκότοπους αλλά είναι συνεχώς δεμένες μέσα στους στάβλους αυτούς. Αναφερθήκαμε επίσης σε μία οδηγία, την 98 58, για την προστασία των ζώων. Σαφώς, η οδηγία αυτή θα πρέπει να βελτιωθεί, αλλά κυρίως θα πρέπει να εφαρμοστεί, να αρχίσει να εφαρμόζεται ορθά αυτή η οδηγία. Αυτό ζητούν και αναφέροντες. Θέλουν στην πράξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να μας δώσει ξεκάθαρες κατευντήριες γραμμές, οι οποίες να πάνε στους εκτροφείς και στους γεωργούς. Όπως ακριβώς έχει γίνει στο παρελθόν και με άλλες διατάξεις, όπως για παράδειγμα η κοπή της σουράς των χείρων ή και σε άλλες περιστάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ χρήσιμη έκκληση που κάνει αυτή η αναφορά και τώρα που ξέρουμε επίση ότι υπάρχει και μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα, ε, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό θεωρώ να αποσταλεί και στην ευρωπαϊκή αυτή πλατφόρμα η αναφορά αυτή, προκειμένου να λάβει γνώση αυτή η πλατφόρμα και προφανώς θα πρέπει να μείνει ανοιχτή θεωρώ αυτή η αναφορά και θα πρέπει να έχουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια έγκριση κατευντήρω γραμμών για την ευζοία των ζώων. Και ξέρετε ότι σε μια πρόσφατη συνεδρίαση της Διακομματικής Ομάδας για την Ευζοία των Ζώων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακριβώς για το ζήτημα αυτό συζητήσαμε, κυρία Πρόεδρε, και ακριβώς θίξαμε ακριβώς τα, τα, τα ίδια ζητήματα σε αυτή τη συνεδρίαση ίδια ζητήματα με αυτά τα οποία μας παρουσίασε ενδιαφέρονται σήμερα. Εν κατακλείδη να πω ότι κατά την άποψή μου το παραγωγικό αυτό μοντέλο το οποίο στοχεύει μόνο στο κέρδος και στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και της παραγωγής δυστυχώς το βλέπουμε πλέον στην Ευρώπη ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο πόρους, σπαταλούμε πόρους ακόμα και στον τομέα αυτό της ε, παραγωγής. Ενώ θα ήταν πολύ πιο σημαντικό, θεωρώ, να αλλάξουμε, αν θέλετε, ρότα και να βρούμε πιο βιώσιμους τρόπους κτηνοτροφίας και παραγωγής που να σέβονται όχι μόνο την ευζοία των ζώων, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει, ιδίως στη χάραξη της μελλοντικής πολιτικής για τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Ελεονόρα. Λοιπόν, Πέτρη Γιάρη, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευημερία, ευζωία των ζώων. Είναι μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία και θεμητή. Τουλάχιστον 20-30 χρόνια μας απασχολεί αυτό το θέμα και θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν και διαφορετικές αντιλήψεις για το τι εστί ευζωία και ευημερία των ζώων και πώς γίνεται αυτή σεβαστή. Είναι το αντιπαράδειγμα στη συνάδελφο Εύη Εγώ θεωρώ ότι η εντατική ε, ε, αγελαδοτροφία που είμαι και αγρότης ε, δεν ανταποκρίνεται σωστά στο είδος των βοηδών. Δεν είναι αξιοπρεπές απέναντι στις απαιτήσεις. Η μικρή η μικρή μικροί κτηνοτρόφη είναι σε καλύτερη μοίρα. Δεν θέλω να σχηματοποιώ τώρα το μεγάλο είναι κακό, το μικρό είναι καλό. Τώρα θα πρότεινα το εξής, να παραμείνει, ε, μάλλον να ε, διαβιβαστεί στο Intergroup για την ευζοία των ζώων αυτή η αναφορά. Ε, έχουμε εδώ δυνάμεις στο Κοινοβούλιο, διακομματική ομάδα το Intergroup αυτό και να περιμένουμε την απάντηση και μετά όταν έχουμε την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουμε για τη μοίρα της αναφοράς αυτή. Δεν έχω κανέναν άλλον στο κατάλογο των ομιλητών. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Όχι. Ωραία. Οπότε, να δώσω και πάρει το λόγο στον κύριο Στίβενσον για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα βοηθούσε να στείλετε την αναφορά στο Intergroup αυτό το έχουν ξαναδεί το θέμα και έχουν εκφράσει και εκείνοι τις ανησυχίες τους για την ευζοία των, αγελδο... των ε, γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Αλλά το Intergroup αυτό δεν έχει τις εξουσίες μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής όπως είναι η δική σας. Και πραγματικά απευθύνω έκκληση να κρατήσετε αυτή την αναφορά ανοιχτή, να κρατήσετε τον έλεγχο και να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές. Οδηγία υπάρχει, είναι καλή οδηγία αλλά εκφράζεται πάρα πολύ γενικόλογα ότι οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να λάβουν όλα τα λογικά μέτρα και τα εύλογα. Ε, χρειάζονται κατευθυντές γραμμές για να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι και τα κράτη-μέλη ποια είναι αυτά τα μέτρα που πρέπει να λάβουν ε, για περιπτώσεις χολότητας, μαστίτιδας, τραυματισμό, ε, τέτοιων νυχτρών, συνθήκων έλλειψη υγιεινής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε εργαστή την περσμένη χρονιά, έβγαλε και έκθεση. Αλλά είναι γελίο να πούμε ότι εδώ σταματάει αυτή η δουλειά και δεν χρειάζεται τίποτα. Η αρχή είναι, όχι το τέλος, για να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε οι γαλακτοπαραγωγές ε, να εκτρέφονται με όρους αξιοπρεπή. αυτό θα πρέπει να ισχύει για κάθε ζώο. Πρέπει, πρέπει να εκτρέφεται υπό αξιοπρεπείς συνθήκες. Αυτό αφορά όλες τις ε, σχετικές αναφορές. Θα ήθελα τώρα να συνοψίσω. Έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες της διακομματικής ομάδας για τα ζώα ε, στο Κοινοβούλιο ξέρουν την κατάσταση, αλλά δεν έχουμε προσπαθήσει ακόμη να διαβιβάσουμε την αναφορά στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας το κάνουμε αυτό, να την υποβάλουμε προς ενημέρωση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και επίσης σκοπό έχω να σας προτείνω να στείλουμε και μία επιστολή στον Επίτροπο Ανδρουεκάητης, επισημένοντας ότι είναι καλή η οδηγία, αλλά δεν εφαρμόζεται πλήρως στα κράτη-μέλη και αν θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο είδους κατευθυντήρια γραμμή, θα ήταν χρήσιμη για να μπορούν τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν ε, βέλτιστες πρακτικές και να μπορούμε μετά βήμα προς βήμα να προχωρήσουμε. Αυτά μπορούμε να κάνουμε για την ώρα και βλέπω ότι γνέφεται καταφατικά και ότι συμφωνείτε μαζί μου. Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ κύριε Στίβενσον γιατί ήσασταν πάρα πολύ θετικός, είναι τόσο ε, καταθλιπτικό το θέμα, αλλά το γεμίσατε με τόσο ελπιδοφόρα μηνύματα για το μέλλον. Ευχαριστούμε λοιπόν, καλά κάνετε και συνεχίστε την καλή δουλειά. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα δούμε τα αποτελέσματα της δουλειάς αυτής. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην Επιτροπή και ε, καλό ταξίδι. Επόμενη αναφορά 0475 εξ ονόματος διαφόρων ενώσεων προστασίας των ζώων ε, ε, φέρουσα 464 υπογραφές σχετικά με την παραμέληση των αδέσποτων ζώων στη Βουλγαρία. Είναι εδώ η αναφέρουσα Μάρτα Γιώργεβα. Καλώς ήρθατε, σας δίνω το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δυστυχώς και άλλες ε, δυσάρεστες εικόνες θα σας δείξουμε. Να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε αυτή την αναφορά εκ μέρους 18 βουλγαρικών ενώσεων προστασίας των ζώων ε, από ολόκληρη τη Βουλγαρία. Εκτιμούμε όλους ιδιαίτερους το ρόλο της Επιτροπής σας ε, στην ε, έγκριση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ε, κατοικιδίων και αδέσποτων ζώων έχουν, ε, έχουμε εκφράσει την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών ε, με τη σημασία ύπαρξης δεσμευτικής νομοθεσίας για την καλύτερο έλεγχο και διαχείριση των αδέσποτων ζώων ε, από την έγκριση του ψηφίσματος το 2012 σήμερα το 2018 όχι μόνο εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα, αλλά έχει επιδεινωθεί και όχι μόνο στη Βουλγαρία, αλλά και σε πολλά ε, κράτη της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, ε, λόγω των εθνικών ε, παραδόσεων στα κράτη-μέλη. Το άρθρο 13 των συνθήκων συστηματικά παραβιάζεται, τη συνθήκη του Άμστερνταμ, που λέει ότι παρέπει τα ζώα να γίνονται σεβαστά κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Η Βουλγαρία ενέκρινε μία ε, πράξη προστασίας των ζώων το 2008. Ε, υπάρχει νομοθεσία που ισχύει από το 2011, η οποία όμως δεν εφαρμόζεται. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το κυβερνητικό, ο κυβερνητικός φορέας που είναι υπεύθυνο ε, για την εφαρμογή, η Υπηρεσία Ασφάλειας των τροφίμων δεν ε, ε, εκπληρώνει τις, ε, δεν σέβεται τις υποχρεώσεις της, τις Στη Βουλγαρία αυτό που αντιμετωπίσουμε είναι παράνομη αναπαραγωγή, πώληση και ιδιοκτησία των ζώων. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ούτε καν ε, για αναγνώριση, ούτε καν ε, για εμβολιασμό κατά της λύσας, για παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλες ανησυχίες για ζητήματα δημόσιας υγείας και κινδύνου όχι μόνο για τους Βούλγαρους βεβαίως. Ε, στα περισσότερα βουλγαρικά σπίτια βλέπετε πώς κρατούνται τα ζώα αυτά με ένα λουρί, δεν, γίνονται, δεν γίνεται κανένα εμβόλιο, με μια αλυσίδα. Ε, υπάρχουν μάλιστα και ιστοτοποί που, δίνουν, που πολλούν ζώα, σκυλιά, ακόμα και για σκυλομαχίες ε, που είναι ένα έγκλημα στη Βουλγαρία, ένα δίκημα. Ε, βλέπετε την κατάσταση στις ε, φωτογραφίες που σας δείχνω. Μία μόνη φορά ε, οι αρχές παρενέβησαν όταν ένα μέλος του κοινοβουλίου σας αντέδρασε αυτά όσον αφορά τα κατοικίδια ζώα. Τώρα, όσον αφορά τα δέσποτα ζώα, σε αυτή την περίπτωση η κακομεταχείριση και η βιαιότητα κατά των ζώων γίνεται από τις τοπικές αρχές, αυτές, τις ίδιες τις τοπικές αρχές, ε, στις ε, ε, δημοτικές εγκαταστάσεις. Είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Χιλιάδες ζώα κρατούνται υπό συνθήκες και πρέπει να ε, μαλώνουν ε, στα κοινοκομεία για την τροφή τους ε, κατά παραβίαση της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων. Δεν την χάνουν δηλαδή, δεν αναλαμβάνονται τα ζώα αυτά από τους υπεύθυνους φορείς. Ε, οι βουλγαρικές αρχές ε, σαμποτάρουν εσκεμένα ε, την νομοθεσία που αφορά την προστασία των αδέσποτων ζώων. Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα, πάρα πολλά χρήματα των φορολογούμενων πηγαίνουν, υποτίθεται, στην βελτίωση των εγκαταστάσεων, αλλά ουσιαστικά είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο βλέπετε μία, ένα από τα εκατοντάδες ε, ε, άλογα που πέθαναν πέρσι στα βουνά εγκαταλελειμμένα. Ε, είχαν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για την αναποραγωγή των συγκεκριμένων, ε, του συγκεκριμένου αλόγου στον ιδιοκτήτη του. Να τι γίνεται όταν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δίνουν, χώρα, δίνουν χρήματα σε μια χώρα που δεν υπάρχει κανένα έλεγχο για την ευημερία των ζώων. Μη κυβερνητικέ οργανώσει και χιλιάδε χιλιάδες άτομα από τη Βουλγαρία και την Ευρώπη έχουν κάνει έκκληση ε, στι βουλγαρικέ αρχέ για να γίνει κάτι. Ε, και στον Εθνικό Συνήγορο του Πολίτη έχουμε ε, κάνει έκκληση. 11.000 υπογραφές εστάλησαν ε, στα αρμόδια Υπουργεία. Μάλιστα υπήρξαν και μερικές υποθέσεις που φτάσαν στη δικαιοσύνη του 2015. Υπήρξε μία απόφαση του Ανώτατου Δικατικού, Διοικητικού Δικαστηρίου, η οποία ακόμη δεν εφαρμόζεται το 2018. Όλα αυτά τα δεδομένα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα σε εθνικό επίπεδο για την υπεράσπιση τη ευημερία των ζώων, ε, την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Σας κάνουμε έκκληση ω Επιτροπή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθήσετε το ζήτημα αυτό και να διατηρήσετε την πίεση στι βουλγαρικές αρχέ για να αναλάβουν δράση για το θέμα αυτό. Κάνουμε έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει την εφαρμογή του ψηφίσματο του Κοινοβουλίου για ένα νομικό πλαίσιο για τα κατοικίδια κατά αδέσποτα ζώα να δει κατά πόσο η Βουλγαρική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων όντως ε, ε, ε, προσπαθεί να επιβάλλει τη σχετική νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή και την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ και τώρα έχει έρθει ώρα να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Το λόγο η κυρία Κούσμα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την αναφέρουσα που ήρθε από τη Βουλγαρία, από ό,τι μαθαίνω, για να παρουσιάσει την αναφορά της. Εγώ τι μπορώ να σας πω. Ότι προσωπικά, πραγματικά έχω συγκλονιστεί από αυτά που μας είπατε, γιατί και αγαπώ τα ζώα και ιδιαίτερα τα σκυλιά και έχω και σκύλο. Αλλά δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτό που είπε και στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς έχει η κατάσταση σήμερα. Δεν υπάρχει νομική βάση για να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευζοία και την ευημερία των αδέσποτων σκύλων, των κατοικιδίων ζώων. Και τα κατοικίδια που ζουν μαζί μας ε, στα σπίτια μας, ε, η ευζοία τους είναι θέμα των κρατών μελών. Υπάρχει μια σύμβαση με το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά αυτό δεν ε, συνιστά ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλούστατα δεν έχει καμία εξουσία και αρμοδιότητα για να ε, παρακολουθεί και να ελέγχει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τη σύμβαση αυτή. Η μόνη δράση που μπορούμε να αναλάβουμε δεν είναι δική μας, είναι δράση των κρατών μελών. Οι εθνικές αρχές μπορούν. Α, και κάτι άλλο που ξέχασα να πω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω συζητήσει, προηγουμένως σας ανέφερα την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ε, που συνεδριάζει την Πέμπτη και σας προσκαλώ να μπείτε στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας αυτής για την ευζοία των ζώων. Βάλτε στο Google EU Platform for Animal Welfare στα αγγλικά. Και θα βρείτε την ιστοσελίδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πλατφόρμα αυτή και το σύνδεσμο ε, στο web streaming και που μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση την 5η 21 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί αρχίζει η συνεδρίαση. Και γιατί τα αναφέρω αυτά, διότι ακόμα και αν δεν έχει ε, καμιά δυνατότητα και καμιά νομική βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα των αδέσποτων σκύλων. Τα μέλη της πλατφόρμας ε, ε θελοντικά δημιούργησαν μια ομάδα που ασχολείται με αυτό το θέμα. Στο διαδίκτυο. Και την Πέμπτη θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της πρώτης του συνεδρίασης. Αυτό ήθελα να σας πω. Και το άλλο Και πάλι στη συνεδρίαση της πλατφόρμας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το πρόγραμμα δράσης της και ελέγχου για την πώληση κατηγηδίων ε, στο διαδίκτυο, γιατί ξέρουμε ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα ε, αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Η Ιντερνετική λοιπόν πώληση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάιτς, πρώτος ε, στον κατάλογο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα τα πω στα αγγλικά. Καταρχάς, δεν ξέρω αν αφήνουν κανέναν εδώ αδιάφορο αυτές οι φωτογραφίες. Και επίσης δεν συμβαίνει μόνο στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία υπάρχουν προβλήματα και στην Ιταλία μεγάλα και αλλού. Και αναφορές από την Ισπανία εξ όσων γνωρίζω. Και καταρχάς θα ήθελα να πιέσω να συλλέξουμε όλες αυτές τις αναφορές που πηγαίνουν στην ίδια κατεύθυνση. Δεύτερον, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. βεβαίω η ευζοία των ζώων δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μπορεί να πιέσει, αλλά μπορεί να πιέσει για τα θέματα δημόσιας υγείας. Και εάν δεν ελέγχεται την αναπαραγωγή των σκύλων και των κατηγιδίων και τη δυνατότητα ε, να τα πουλάει ο καθένας όπου θέλει, τότε τελικά αυτό είναι εις βάρος της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μοχλός πίεσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, από όλο αυτό το παράνομο εμπόριο και την αναπαραγωγή έχουμε και λαθρεμπόριο ε, ζώων που περνούν τα σύνορα και τα πουλούν τα ζώα αυτά στην ε, Αυστρία, τη Γερμανία που ο κόσμος αγαπάει τα ζώα και είναι πρόθυμος να βάλει και βαθιά το χέρι στη τσέπη. Πρόκειται και για διασυνεριακό λάθρεμπόριο ζώων. Και τελικά ποιο ε, είναι το αποτέλεσμα ότι υπάρχει πολύ αυστηρή νομοθεσία για την αναπαραγωγή Γιατί αν έχετε πολύ αυστηρή νομοθεσία με ένα τσιπάκι ε, που ε, βλέπεις πώς έγινε η παραγωγή, ποιοι είναι οι γονείς του, πώς ε, έχει γεννηθεί και πού το ζώο και μπορείς όλα αυτά να τα αντιμετωπίσεις, να τα ταυτοποιήσεις και άμα το βρεις αυτό το ζώο αδέσποτο υπάρχουν και νομικές συνέπειες. Λοιπόν, να μην παραμείνει απλώ ανοιχτή αυτή η αναφορά, να συνδεθεί και με όλε τι υπόλοιπε που πηγαίνουν προ την ίδια κατεύθυνση. Και προηγουμένω μιλήσαμε και για ένα άλλο θέμα ευζοίας των ζώων, το ξέρω ότι δεν θα ληφθούν νομικές αποφάσεις για αυτό το θέμα ε, στην πλατφόρμα και στο Intergroup είναι ότι εδώ στο Intergroup έχουμε ε, διακομματική ομάδα, είναι πολλές πολιτικές ομάδες σχεδόν και ενώνουν τις δυνάμεις τους για να υπερασπιστούν την ευζοία των ζώων. Και αν υπάρχει ψήφισμα ή μια δυνατότητα να αρχίσει μια νομική διαδικασία να το ε, ξαναβάλουμε και να έχουμε μια καλή αρχή ε, στο Intergroup. Προηγουμένως ακούσαμε για τις αγελάδες και πρόσφατα Έχουμε συζητήσει στο Intergroup το θέμα των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων, αλλά έχει το θέμα των κατοικιδίων. Παρακαλώ λοιπόν να διαβεβαστεί αυτή η αναφορά στο Intergroup για την ευζοία των ζώων για να αρχίσει μια διαδικασία για ένα νέο ψήφισμα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν σα δώσω το λόγο κύριε Μαλίνοφ, εμείς δεν μπορούμε να αρχίσουμε νομικές δράσεις εξ ονόμα της Επιτροπής μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κάνει αυτά. Εμείς δεν έχουμε καμία εξουσία προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, εσείς κύριε Μαλίνοφ. Ε, δεν είναι και οι καλύτερε ημέρε αυτέ για του βουλγάρους Ευρωβουλευτέ, όλα αυτά που συζητάμε στην Επιτροπή μα. Διάβασα την αφορά αυτή το πρωί Μάλλον το πρωί ασχοληθήκαμε με μία αναφορά την οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι βούλγαροι πολίτες, ενώ τώρα ασχοληθήκαμε με μία αναφορά η οποία είναι πιο κρυφή αν θέλετε. Δεν έχει τέτοια προβολή, αλλά είναι εξίσου δυνηρή. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση αυτή, μας διανεμήθηκε μία δήλωση από την Διακομματική Ομάδα για την Ευζοία των Ζώων, η οποία συνδέεται άμεσα τα όσα συζητάμε και μάλιστα αναφέρεται ρητά στην ε, αναφορά αυτή που συζητάμε τώρα. Και το Intergroup αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2012 όταν ε, η τότε αναφορά ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει δράση. Και γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκτοτε δεν έχει υποβάλει καμία νομοθετική πρόταση για την προστασία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων μολονότι υπάρχει πολιτική βούληση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί δεν μπορούμε να αναλάβουμε νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά υπάρχει μια ειδική δήλωση δικιά μα από το Intergroup. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι και αυτή η αναφορά για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα νομικό κενό στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλώντας εξ ονόματος και του ΕΛΚΑ θα έλεγα ότι α, τα όσα ακούσαμε αυτή τη στιγμή συνάδουν απόλυτα με αυτά τα οποία πιστεύω εγώ σαφώ δεν θα πρέπει να πούμε στου Ευρωπαίου πολίτε, αυτά που μόλι τώρα μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ήρθε και μα είπε τεράστιο το πρόβλημα, συμφωνούμε μαζί σα, δεν υπάρχει νομική βάση, κλείνει η αναφορά. Ε, Ακριβώ αυτό δεν πρέπει να το πούμε σε κανένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω στου Ευρωπαίου εκείνου πολίτε οι οποίοι κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια για να έρθουν εδώ και να παρουσιάσουν την υπόθεσή του στην Επιτροπή μα. Λοιπόν, τι έχω να προτείνω. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Γνωρίζω ότι δεν έχουμε ούτε τους πόρους, ούτε το χρόνο για να πάμε στη Βουλγαρία μέσω μιας αποστολής. Πάντως θα ήθελα να διοργανωθεί μη τι άλλο μία αποστολή και να μπορέσουμε στην αποστολή αυτή να φέρουμε και συναδέλφους από το Intergroup, από τη διακομματική ομάδα. Ξέρω ότι δεν θα είναι επίσημη αυτή η αποστολή, αλλά ξέρετε μερικέ φορέ οι ανεπίσημες επισκέψεις έχουν μεγαλύτερη επιρροή από τι επίσημες. Επίσης, να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει ήδη ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου από το 2012. Και μια άλλη πρόταση που θα ήθελα να κάνω και που συνδέεται με την κατάσταση την οποία συζητάμε τώρα, θα ζητούσα ή δυνατόν, αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το ζήτημα αυτό, ας μην πει Σόνη και καλά ότι πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά, γιατί αν χρειαστεί να ψηφίσουμε και δεν έχουμε ε, απαρτία, αυτό θα είναι ιδιαίτερα υποτιμητικό θεωρώ για όλου μα και απαξιωτικό για όλου μα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και σαφώ θα πρέπει ομόφωνα να υποστηρίξει την επίλυσή του η Επιτροπή μα. Ε, ας το πετύχουμε αυτό, ας κρατήσουμε αν μη τι άλλο ανοιχτή την αναφορά και στο το πετύσουμε αυτό ομόφωνα προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και εμείς να βοηθούμε τους αναφέροντες στον αγώνα τους αυτό. Πρόεδρος, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο μου ζητάτε. Αυτή η ομοφωνία την θέλω εγώ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε αυτή την ομοφωνία πιο συχνά, θα διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή μου. Ο κύριος Πυρίνσκι τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι οι αναφέροντες απευθύνονται εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη δική μας την Επιτροπή, έχοντας προφανώς εξαντλήσει κάθε δυνατό διάβλο που είχαν ε, σε εθνικό επίπεδο για το πολύ δύσκολο αυτό πρόβλημα. Και βέβαια έχουν απευθυνθεί σε όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό. Θλιβερό ακριβώς επειδή ε, είναι προφανής η σοβαρότητα της κατάστασης και συγκλονίσει τους πάντες. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή μας. Ποια θα αρέσουμε ότι θα είναι η δέουσα λύση εδώ πέρα. Οι αναφέροντες έχουν κάνει δύο εκκλήσεις αν θέλετε. Πρώτον, ζητούν από την Επιτροπή μας να συζητήσει προφανώς αυτήν την αφορά, αυτό το κάνουμε τώρα. Και η δεύτερη έκκληση των αναφερόντων έχει να κάνει με μία επιτόπου εξέταση και αξιολόγηση των προβλημάτων που περιγράφουν και γίνεται μία έκκληση για την διοργάνωση διερευνητικής απόστολης. Κύριε Μαλίνοφ, εσύ μας είπατε ότι ενδεχομένω να πάτε και μόνος σας επιτόπου ή να συστήσετε μόνος σας μια τέτοια ομάδα άτυπη για να πάει στη Βουλγαρία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία αυτή του κυρίου Μαλίνοφ και να καλέσουμε όσους παίρνουν το λόγο και ενδιαφέρονται για το ζήτημα αυτό να συμμετάσχουν σε μια τέτοια αποστολή. Αναγνωρίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι σαφώς μόνο βουλγαρικό, ξεπερνά τα σύνορα της Βουλγαρίας, αλλά ότι παρουσιάζεται με μεγάλη σοβαρότητα και σε μεγάλη έκταση στη χώρα αυτή. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2012 για αυτό το ζήτημα, στο ψήφισμα αυτό καλούμε καταρχάς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να επικυρώσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά και να μεταφέρουν τι διατάξει σύμβαση αυτή στην Εθνική Νομοθεσία και καλεί, κατά δεύτερο λόγο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία των αδέσποτων και των ζώων συντροφιά, όπου να περιλαμβάνονται και κανόνε για τον εντοπισμό και την καταχώρηση των ζώων. Υπάρχουν συγκεκριμένε στρατηγικέ για τα δέσποτα ζώα, όπω για παράδειγμα στήρωση και εμβολιασμό, μέτρα στον αφορά την πρόθεση τη υπεύθυνη ιδιοκτησία των ζώων αυτών, υπάρχουν τα απαραίτητα καταφύγια για τα ζώα αυτά, καθώς επίσης και οι απαραίτητες διατάξεις όσον αφορά το, την αντιμετώπιση των δέσποτων ζώων και επίση να υπάρχουν συγκεκριμένε αυστηρέ κυρώσει για οποιοδήποτε κράτο μέλο δεν συμμορφώνεται με αυτού του κανόνε. Και μετά από όλα αυτά που ζητά το ψήφισμά μα, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μα λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν δίνεται να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ζητήματα αυτά. Μα αυτό είναι απίστευτο. Απίστευτο. Και όπως είπε ο κύριος Μαλίνοφ, πραγματικά αυτό δείχνει πλήρη απουσία ανάληψης ευθύνης. Και δεν θα ήθελα να τα πω τα πράγματα με πιο αυστηρό τρόπο. Σαφώς θα πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτή την αναφορά και ας δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε αρμοδιότητα έχουμε που έχει η Επιτροπή μας και εν το Κοινοβούλιο προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε μη τι άλλο κάποια θετικά αποτελέσματα σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό που είπατε, αυτό που παραθέσατε είναι τμήμα της δήλωσης ε, της ε, διακομματικής ομάδας ε, που το λάβαμε μόλις σήμερα. Η κυρία Εύε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που ακούω πολλούς συναδέλφους οι οποίοι στηρίζουν αυτή την αφορά γιατί επιτέλους το θέμα αυτό λαμβάνει τη δέουσα προσοχή Πάρα πολλές αναφορές είχαμε στο παρελθόν για το ζήτημα αυτό, τις οποίες τις κλείσαμε εξαιτία της αρνητικής απάντησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μας έλεγε πάντοτε δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο, νομική βάση για να αναλάβει δράση, δεν υπήρχε κοινοτική νομοθεσία για αυτό το ζήτημα. Πάρα πολλέ αναφορέ όμω λάβαμε στην Επιτροπή μα τελευταία χρόνια, οι οποίε κλείσανε. Επιτέλου φαίνεται ότι υπάρχει ένα κάποιο άνοιγμα, ότι κάτι διαφορετικό ενδεχομένω να προκύψει και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω μια τέτοια θετική ανταπόκριση από τους συναδέλφους. Νομίζω ότι έχει το πλήρωμα του χρόνου και δεν επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, να πιέσουμε περισσότερο σε Επιτροπή Αναφορών. Έχουμε πλέον συγκεκριμένες μελέτες, από το Policy Department έχει γίνει μάλιστα μια μελέτη, εμείς τη ζητήσαμε ως Επιτροπή Αναφορών, και βλέπουμε ότι στη μελέτη αυτή υπάρχουν συγκεκριμένα πλέον πορίσματα όσον αφορά το ζήτημα αυτό για τα ζώα συντροφιά και τα δέσποτα ζώα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα και θα πρέπει επιτέλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλη νομοθετική πρόταση. Α μην ξεχνάμε πόσε δυσκολίε εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο σε πάρα πολλέ χώρε γύρω από το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι πλέον η λύση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ πολύ. Όπως βλέπετε κυρία Γεωργίευα, υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη των ε, επιχειρημάτων σας και ολόκληρης κατάστασης ε, που μας ε, παρουσιάσατε και προφορικά αλλά και μέσω πολύ έντονων φωτογραφιών. Θέλετε να πάρετε και πάλι το λόγο. Ναι, Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους ε, τους ευρωβουλευτές ε, για ε, την έκφραση της άποψής σας. Εμάς πραγματικά μας αγγίζει αυτό. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπουν οι κανόνες, να δώσω στην κυρία Παπαδόποβα το λόγο να πει έστω και μία πρόταση στα βουλγαρικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω πολύ και να πω ότι αυτό το πρόβλημα αλήθεια ε, ε, είναι πραγματικό και σημαντικό. Δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Ε, δεν είναι απλώς μια προειδοποίηση το πρόβλημα των αδεσπότων ε, σκύλων αφορά ε, την υγεία των Ευρωπαίων και τα συναισθήματα των Ευρωπαίων. Αυτά που σας δείξαμε εδώ, οι φωτογραφίες από τις αυλές και τους δρόμους στη Βουλγαρία ε, είναι κάτι το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την παράκληση να κάνει κάτι. Και όταν παίρνετε αποφάσεις σκέφτεστε αυτό, που σας είπαμε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να συνοψίσω. Πρώτον, θα πρέπει να στείλουμε επιστολή ε, στον Επίτροπο της και για αυτό το θέμα. Α, δεν ε, σας είχα δει, δεν είχα ζητήσει προηγουμένως το λόγο κύριε Έκα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη. Θα μιλήσω γερμανικά. ο συνάδελφος Μαλίνοφ είχε μια πολύ καλή ιδέα. Να πάμε στη Βουλγαρία, να δούμε τι γίνεται επί τόπου, η ερευνητική αποστολή, για να κοιτάξει τα πράγματα επί τόπου. Και έτσι πολύ αυθόρμητα ε, του προτείνω την υποστήριξή μου. Έχω πάει πέντε φορές στη Ρουμανία. Ε, είμαι ειδικό πλέον στα αδέσποτα. Ε, ο κύριος Πανσέσκου μετά που πήγα εγώ τόσες φορές, στο ίδιο το κοινοβούλιο κατέβηκε, στο, στην τοπική βουλή ε, του Βουκουρεστίου, χρειάστηκε να φύγει από τη χώρα. Και ο ίδιος ο δήμαρχος του Βουκουρεστίου, δεν ξέρω, μπορεί να βοήθησα κι εγώ λίγο. Και μετά από 1,5 μήνα τον καθαίρεσαν και τον φυλάκισαν. Λοιπόν, να οργανώσουμε κάτι με τους συναδέλφους για να πάμε στη Βουλγαρία και να κάνουμε κάτι για αυτά τα δέσποτα ζώα. Ευχαριστώ. Okay, we are not talking about... Ωραία. Τώρα μιλάμε για τη Βουλγαρία, έτσι. Ναι, ναι, για τη Βουλγαρία, για τα δέσποτα ζώα στη Βουλγαρία, για τα σκυλιά. Ξέρουμε ότι συμβαίνουν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια φρικτά φαινόμενα, αλλά ας παραμείνουμε στο θέμα μας που είναι η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εάν το επιθυμούν οι συνάδελφοι, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες και το ΕΛΚ ζητούν να πάμε αποστολή ε, στη Βουλγαρία. Πείτε το στους συντονιστές, εάν το θέλουν και οι δύο, ήδη έχουμε επιτροπή, ε, πλειοψηφία στην Επιτροπή μας. Οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ, αν το φέρουν ε, στους συντονιστές, θα εγγραφεί στον κατάλογο για την επόμενη χρονιά πλέον όμως αυτό είναι πολύ πιο ισχυρό από ότι μια μονομελής αποστολή. Κύριε Μαλίνοφ, ξέρω ότι είστε πολύ ισχυρός ανήρ, αλλά εάν ε, μπορούμε να πάμε κανονική αποστολή και να κάνουμε συστάσεις και έκθεση, αυτό μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Λοιπόν, αν αποφασίσει η Επιτροπή, να ε, το συζητήσουμε στους συντονιστές και νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Και όπως σας είπα, έχετε ήδη την πλειοψηφία σοσιαλιστέ και δημοκράτε. και ελκύστε οι δύο μεγαλύτερε ομάδε. Λοιπόν, θα στείλουμε και επιστολή στον Επίτροπο Ανδροϊκάητη για το θέμα αυτό, όπω και για το προηγούμενο. Και να το παραπέμψουμε και στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μάθαμε τώρα ότι υπάρχει, διότι προφανώς το Intergroup για την ευημερία των ζώων στο Κοινοβούλιο έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες θα επανέλθω όμως σε αυτό που μας είπανε στη δήλωσή τους, ότι θα ήθελαν το Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε μια συνεδρία ενδιαφερομένων για να αποτιμήσει την κατάσταση ξανά και να προσπαθήσει να βρει λύσεις. Είναι πολύ καλές αυτές οι προσπάθειες λοιπόν που γίνονται από το Intergroup για να πούν ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Άρα να του στείλουμε την ενημέρωση για το τι θα κάνουμε με αυτή την αναφορά για να είναι και αυτοί ενήμεροι και να συμμετέχουν. Α, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, επιστολή στο βουλγαρικό οργανισμό ασφάλειας τροφίμων που υπάγεται στο αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας Τροφίμων και Δασών. Το 2017 τον Ιούλιο έστειλαν μια απάντηση στην Επιτροπή μας και είπαν ότι το πρόβλημα με την προστασία των αδεσπότων ζώων είναι υψής της σημασίας. Οπότε τι κάνανε έκτοτε λοιπόν αφού μας στείλαν αυτή την επιστολή ότι είναι τόσο σπουδαίο το πρόβλημα αυτό. Θα πιέσουμε να μας πούνε τι συγκεκριμένα μέτρα έλαβαν ή δεν έλαβαν. Μπορεί να το ξέχασαν κιόλας, ποιος ξέρει. Καμία παράληψη. Ε, αυτά μπορούμε να κάνουμε εμείς στην παρούσα στιγμή. Λοιπόν, συμφωνείτε όλοι να προχωρήσουμε έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ. Έτσι θα προχωρήσουμε. Και ας προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη αναφορά υπαριθμών 720. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, να πω σε όλους τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στις Βρυξέλλες και για όλες τις προσπάθειες που κάνετε και έχετε κάνει επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια σε τόσο διαφορετικά φόρα. Σας ευχαριστώ και πάλι και καλή επανόδο στη χώρα σας. Item 20. Είναι το σημείο 26 σχετικά με την ε, κατάσταση των γυναικών που κρατούνται παρά τη θέλησή τους σε καταβλισμούς Σαχράουι στο Τιντούφ της Αλγερίας. Η Μαρία Ελίσσα Παβών Μουλέρο παρευρίσκεται η αναφέρουσα και με χαρά τη δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Λέγομαι Λίσα Παβών και έρχομαι εδώ εκπροσωπώντας πολίτες για την ναι, οργάνωση «Η ελευθερία είναι το δικαίωμά τους». 50 γυναίκες έχουμε φιλοξενήσει, ενήλικες, Σαχράουι, που τις ε, κρατούν εχμάλωτες παρά τη θέλησή τους στους καταβλισμούς των Σαχράουι στην Τιντούφ έχουμε ανάδοχες οικογένειες και οικογένειες που έχουν υιοθετήσει, τέσσερις ε, που με συνοδεύουν οι πατέρες και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας εξηγήσω το πρόβλημα και να σας ζητήσω να μεσολαβήσετε για να φεθούν ελεύθερες όλες αυτές οι γυναίκες για να επιλέγουν τι θα κάνουν στη ζωή τους ασκώντας ε, το δικαίωμα σε αυτό εκτός των καταβλισμών έχουμε την παρουσίασή μας με φωτογραφίες από διάφορες γυναίκες, Μαλώμα, Κορία, ε, Ντάρια και Μαγίμα, για να δείτε πώς παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι ε, κρύβει το μέτωπο πολυσάριο και το περιβάλλον τους, γιατί επικαλείται το πολιτισμό και ε, την ε, παράδοση. Είναι ενήλικες που τις κρατάνε οι εχμάλωτες, ομήρους είναι βία, έμφυλη αυτή εις βάρος των γυναικών. Είναι ενήλικες και παρόλα αυτά οι οικογένειές τους τους επιβάλλουν μια ζωή που δεν έχουν επιλέξει με σωματική και ψυχική κακοποίηση, με αναγκαστικές ε, γάμους με το στανιό για να γίνουν μητέρες ε, έχουν έρθει στην Ισπανία γύρω στο 2000 ως παιδιά για διακοπές και παρέμειναν για λόγους ιατρικούς ή μετά από απόφαση των βιολογικών τους γονέων που θέλησαν να τους δώσουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον. Ωστόσο, όταν ε, ενηλικιώθηκαν, οι βιολογικές τους οικογένειες ε, θεώρησαν ότι είναι κτήμα τους. Αυτό είναι δικαίωμα απαράδεκτο, ε, ανύπαρκτο και παράνομο. Και είναι τελείως φαλοκρατική αυτή η μορφή κοινωνίας, ε, πατριαρχική, φιλετική και ακραία. Το μέτωπο Πολυσάριο που κάνει κομμάντο στους καταβλισμούς δεν ανταποκρίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, στα εδάφη που ελέγχει. Επιτρέπει και δικαιολογεί αυτά τα αδικήματα, αυτά τα εγκλήματα που είναι τελείως ε, ατιμόρυτα και ποινικοποιεί μάλιστα τα θύματα και τις οικογένειες που τους υποδέχονται στην Ισπανία. Η οργάνωσή μας έχει καταγγείλει το μέτωπο Πολυσάριο για συνενοχή και διαπλοκή για ε, ε, κρατήσεις αυθαίρετες και ε, με τέσσερις ε, περιπτώσεις και τέσσερις συγκεκριμένες καταγγελίες. Το Μάρτιο του 2017 έχουν δρομολογηθεί αυτές. Και τα θύματα, οι γυναίκες αυτές αποκαλύπτονται και ζητούν τη βοήθεια για να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιες για τη ζωή τους. Όσο όμω βρίσκονται στους καταβλισμού, αυτό δεν είναι δυνατό. Η οικογένεια, οι φίλοι και η κοινωνία ασκούν αφόρητε συστηματικές πιέσεις στις γυναίκε αυτέ. και αυτό είναι μια διαρκής ψυχολογική κακοποίηση που τις γονατίζει και πολλές φορές θέλουν και να αυτοκτονήσουν γιατί προτιμούν να πεθάνουν παρά να ζουν τέτοια ζωή όπως το έκανε ήδη η Μαλώμα. 50 τέτοιες περιπτώσεις έχουμε σημειώσει. Τέσσερις όμως ε, δημοσιοποιούμε γιατί οι υπόλοιπε φοβούνται. Οι δύο είναι Ισπανίδες ε, πολίτες που τις έχουν ε, απαγάγει διάφορα μέλη της οικογένειάς τους, τις βάλανε με το ζόρι σε αυτοκίνητο, ε, ξυλοκοπώντας τις, με καταναγκαστική ε, παντριά. Δυόμιση χρόνια κρατάνε μια γυναίκα 25 χρονών και μια άλλη 27 ετών πάνω από 7 χρόνια την κρατάνε τελείως απομονημένη, χωρίς να επικοινωνεί στην έρημο με βαριά ε, ε, ασθένεια που έχει στην καρδιά της και κινδυνεύει η ζωή της. Πέντε τέτοιες περιπτώσεις Ισπανών πολιτών, ανδρών και γυναικών ενηλίκων ξέρουμε τα τελευταία χρόνια και σήμερα υπάρχουν και περισσότερες. Άλλη μία. Άσμα λέγεται και είναι η κόρη της Μαλώμα καρπός ε, ανακαστικού γάμου πέντε μηνών μόνο. Οι άλλε νέε που βλέπετε ε, διαμένουν ε, μόνιμα στην Ισπανία και ε, με το ζόρι τη κρατάνε τέσσερα χρόνια χωρί χαρτιά. 27 ετών και 26 δύο γυναίκες είπαν στο Human Rights Watch, στο παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων θέλουν να γυρίσουν στην Ισπανία. Αλλά η Μαλώμα είναι κόρη μιας βουλευτίνας του μετόπου Πολυσάριο που δεν θέλει να την αφήσει να ζήσει ελεύθερη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει υπέρ των γυναικών αυτών και η, υπηρεσία Ευρωπαϊκής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ε, λάβει εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε το μέτωπο Πολυσάριο, ε, η αλγερινή κυβέρνηση που διαχειρίζεται αυτούς τους καταβλισμούς και η ισπανική κυβέρνηση να εγγυηθούν ε, τα δικαιώματα των τεσσάρων αυτών γυναικών και των υπολείπων να αφαιθούν ελεύθερες και να μπορούν να ζουν ελεύθερα εκτός των καταβλισμών. Θέλουμε να σας ζητήσουμε ρητά να μεσολαβήσετε έτσι ώστε να επιτύχουμε την άμεση επέμβαση της ΥΠΑ της εκπροσώπου ε, Φεντερίκα Μογκερίνη. δεν ξέρω πώς να μεσολαβήσετε και με ποιον έτσι ώστε η Ισπανική κυβέρνηση να μπορέσει να αναγνωρίσει και να καταγράψει επίσημα ε, την κόρη της Μαλώμα ως ε, Ισπανίδα πολίτη και ε, Ευρωπαία πολίτη, αυτό το κοριτσάκι των πέντε μηνών, αυτό το βρέφος. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και για την υποστήριξή σας. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μάλλον ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης δεν έχω το όνομά σας, πάντως έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα τα πω στα αγγλικά. Πράγματι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ε, ε, της οποίας ηγείται η Φεντερίτα Μογκερίνη, ε, προσπάθησε και στις Βρυξέλλες και ε, στις αντιπροσωπείες μας στην Αλγερία να θέσει το θέμα. Είναι ένα ζήτημα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει να κάνει βέβαια και παράλληλα με τα δικαιώματα των γυναικών. Ε, κάτι το οποίο επίσης προσδίδει μια άλλη σημαντική πτυχή ε, υπάρχει και η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συστάσεις της ε, και όλα αυτά τα οποία μας είπατε, τα διαβάσαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουμε καμία ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών η οποία να λέει ότι το ε, Πολυσάριο έχει κάποια ενεργό συμμετοχή σε, αυτές τις, σε αυτά τα περιοριστικά μέτρα κατά των νέων αυτών γυναικών εκτός δηλαδή από τις ε, οικογένειές τους. Παρόλα αυτά, το εξετάζουμε αυτό το θέμα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ήδη κάποιο είδους ε, διαμεσολάβηση ε, μεταξύ πολλών ε, μερών, ενδεχομένως όχι λόγω της καταχώρηση τη άσμα ως Ισπανίδας πολίτη, αλλά εν πάση περιπτώσει το δικαίωμά τους να διαλέξουν που μπορούν να μείνουν. Θα το παρακολουθήσουμε πάντω το ζήτημα αυτό Προφανώ χρήζει μια συντονισμένη προσέγγιση με την Ισπανία που είναι ε, βέβαια υπεύθυνη όσον αφορά την προξενική διάσταση και θα παραμείνουμε πολύ προσεκτικοί, ειδικότερα στο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είπατε κι εσείς και στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας προετοιμασία ε, και εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταβλισμού στην Τουφ της Αλγερίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ ποιος θέλει να πάρει το λόγο, η κυρία Εσταράς. Πρώτη κυρία Πεσέρα, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες ε, που ήρθαν για να μας παρουσιάσουν έναν τρόπο τόσο συγκλονιστικό, όχι μόνο τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά, αλλά και τον πόνο, το γολγοθά όλο αυτό που έχουν ζήσει και την έλλειψη απάντησης στις γυναίκες αυτές. Χαίρομαι πολύ που ακούω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για της αντιπροσώπου της. Πραγματικά πρέπει να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και να αναζητήσουμε ενεργά λύσεις. Περί αυτού πρόκειται. Θα ήθελα λίγο να επιμείνω στο εξή. Ευθύνη φέρει και το μέτωπο Πολυσάριο από τη Σκοπιά τις δράσεις που θέλουν να έχουν και αποκαλούνται να έχουν. Έχουν αυτό η κυβέρνηση ε, της ε, αραβικής δημοκρατίας των Σαχράουι. Ε, υποτίθεται ότι κυβερνάνε και στους καταβλισμούς. Δεν μπορούν να κρατούνται οι γυναίκες παρά τη θέλησή τους. Και το μέτωπο Πολυσάριο ως συνομιλητής και ως ε, συνεργά της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει και ενίσχυση οικονομική. Και γι' αυτό θέλει να αναγνωριστεί ως διεθνής παράγων. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Πολυσάριο όταν λέει ότι δεν μπορεί να λύσει ένα τέτοιο πρόβλημα παράνομης κράτησης γυναικών στους καταβλισμούς που σε πολλές περιπτώσεις έχουν δηλώσει ρητά την πρόθεσή τους να ε, επιστρέψουν στα μέρη από που... Δεν υπάρχει καμία παράδοση, κανένα έθιμο φιλετικό που να κυριαρχεί επί των διεθνών συμβάσεων και των υποχρεώσεων που έχουμε. Και σε αυτό όλοι συμφωνούμε. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι πρέπει να σεβόμαστε παραδόσεις όπως είναι ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ή το δικαίωμα κάποιων οικογενειών να παντρεύουν με το ζόρι τα παιδιά τους. Αυτό λοιπόν επειδή το έχουμε λιμένο και επειδή ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε προσυπογράψει την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι το νομικό πλαίσιο το αντίστοιχο, θα πρέπει να έχουμε και ανάλογη συμπεριφορά εδώ και δράση. Και πέρα από την έκκληση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία και ευχαριστώ, επιβεβαιώνει ότι είναι γνώση της όλα αυτά και είναι έτοιμα τα μέτρα για να δράσουν. Θέλω όμως και η Επιτροπή μας να απευθύνει έκκληση στην Ισπανική κυβέρνηση τώρα, ε, για να συμμετέχει. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που είναι η καινούργια κυβέρνηση, έτσι ώστε Πρώτον, να πολιτογραφήσει ε, η ε, αυτό το κοριτσάκι, το, το πεντάμινο, γιατί είναι κόρη Ισπανίδας. Και ε, μας υποχρεώνει γι' αυτό και η Ισπανική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ισχυρισμού ότι οι βιολογικέ οικογένειε έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν με τα κορίτσια του, με τα παιδιά του, γιατί λέει είναι Πρόκειται για γυναίκε, ε, ε, και δεν είναι μόνο αυτέ οι περιπτώσει, που είναι παρόντες εδώ οι γονείς, μιλάμε για 50 γυναίκες. Δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι ένα μοντέλο αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να δράσουμε. Και πραγματικά προσβλέπω στην Επιτροπή μας για να κάνουμε κρούση στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα αλλά και στην Ισπανική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. you very Ευχαριστώ πολύ, κυρία Εσταράς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνο με την Πεατρίθ Μεσέρα, Ευχαριστώ τους αναφέροντες ε, που ήρθαν μέχρι εδώ και την Ελίσσα Παβών και τις τέσσερις οικογένειες που είναι εδώ παρούσες. Το θέμα πραγματικά αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του για διάφορους λόγους. Σήμερα πρόκειται για τέσσερις οικογένειες. Τέσσερις οικογένειες που ε, ήταν, είχαν ανάδοχες οικογένειες, υιοθεσίες ε, στις ε, διακοπές φιλοξενούσαν αυτά τα παιδιά, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μαζί τους ανάδοχοι γονείς που είχαν και μόνιμη επαφή με τους βιολογικούς γονείς και σε πολλές περιπτώσεις ε, πλήρωσαν και κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις και έσωσαν ε, τις ε, τη ζωή μιας κοπέλας που είχε πολύ σοβαρά προβλήματα και χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Ήταν πάντα στον πλευρό αυτό το κορισιόν και μετά τη στιγμή που ενηλικιώνονται κάποια στιγμή γυρνάνε στους καταβλισμούς οι γυναίκες αυτές. Πολύ ωραία τα είπε η Μπεατρίθ και τους παραβιάζουν απολύτως και τα γυναικεία τους και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τους στερούν την ελευθερία τους δια της βίας και κινδυνεύουν και σωματικά και ψυχολογικά και κινδυνεύει η ακαιρεότητά τους, η σωματική. Υποτίθεται ότι είναι οικογένεια και ε, τα ενίκουμε ή δήμο σε καμία περίπτωση. Ε, ε, όλοι μας θα πρέπει να αντισταθούμε. Και παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας, της αξιοπρέπειας και της ίδιας της δικαιοσύνης. Τους κρατάνε τα διαβατήρια. Όταν σου παίρνουν τα χαρτιά στη μέση της ερήμου, την άδεια παραμονής, το διαβατήριο αυτό είναι απαγωγή κανονική και εχμαλωσία, γιατί ε, εξολοθρεύεται η ελευθερία σου και είσαι κρατούμενη πραγματικά και αναγκάζονται να ε, απεμπολίσουν την ελευθερία τους και ε, οποιασδήποτε προοπτικές για τη ζωή του. Και μάλιστα και τις θεραπείες τους, γιατί μια από αυτές τις γυναίκες κινδυνεύει, κινδυνεύει η ζωή της και τις απομακρύνουν από ένα ασφαλές περιβάλλον που θα μπορούσαν να επιλέξουν αν ήταν ελεύθερες. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, φυσικά δεν έχουν κοινωνικά δικαιώματα, ούτε ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας, ούτε ελευθερία τελεία. Οπότε, όλες οι οικογένειες απευθύνθηκαν στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και ο Γενικός Γραμματέας Ban τότε, το 2017, ασχολήθηκε με το θέμα αυτό για την Τάρια, την Ατζίβα και την Μαλώμα και είπε ότι είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στην ετήσια έκθεση του Συμβούλιο Ασφαλείας για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα ασχολείται με αυτές τις τρεις νέες που κρατούνται παρά τη θέλησή τους. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία στην Επιτροπή μας να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε βραβευθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρηνή και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας θα είναι πάντα απέναντι στην αδικία και στο πλευρό του αναφέροντος ε, όταν παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Και αυτή η περίπτωση τέτοια είναι και μπορούμε να πιέσουμε και να βοηθήσουμε όχι μόνο τις τέσσερις οικογένειες και ε, τις θαραλέες οικογένειες που είναι εδώ παρούσες αλλά και τις άλλες πολύ περισσότερες έτσι ώστε κυρίως να αποτρέψουμε στο μέλλον οικογένειες αυτές που είναι ανάδοχες και είναι πάρα πολλές να μην του συμβεί κάτι τέτοιο. Σήμερα με πήρε το μεσημέρι ένας ε, φίλος μου από την Ιμπίθα και ε, έχει έναν ανάδοχο τέτοιο κοριτσάκι και λέει τι θα γίνει τώρα στο μέλλον θα μου συμβεί και εμένα το ίδιο ίδιες οικογένειε θα λένε αυτά και η Μπεατρίθ η κυρία Μογκερίνη να επιληφθεί ως ύπατη εκπρόσωπος για τα εξωτερικά θέματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει ε, διάβημα στην Ισπανική κυβέρνηση για να ανοίξει τα χαρτιά της και να αναλάβει δράση. Η νέα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που ε, ε, είναι αρμόδια για τα δικαιώματα ισότητας και έχει και δικαιοδοσία απέναντι στους άλλους υπουργούς να αναλάβει δράση. Και το κάνουν ακριβώς με τις γυναίκες αυτό. Γιατί θεωρεί το πολυσάριο ότι ο άνδρας έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου στη γυναίκα. Και επιπλέον η Ισπανική κυβέρνηση να ειδοποιηθεί και η κυβέρνηση της Αλγερίας, ε, ε, το Πολυσάριο, είπατε εκπρόσωπος, γιατί η αλγερινή κυβέρνηση έχει ε, εμπλοκή στην μεταφορά των γυναικών αυτών, πώς πηγαίνουν μέχρι εκεί. Και η Επιτροπή Ντροά, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να ασχοληθεί το θέμα αυτό και η Επιτροπή Εξωτερικών. Για να πιέσουμε να λυθεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Mr. Ευχαριστώ κύριο Γιάρ. Πάρα πολύ σύντομα να συμπληρώσω κάτι. Αν κατάλαβα καλά, για να καταλάβουμε, είναι Ισπανίδες, έχουν ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Φανταστείτε μας πάρουν εμάς τους τέσσερις. Εμείς τέσσερις εδώ, πέντε πόσοι είμαστε. Για ελάτε να πάμε στο Τιντούφ λοιπόν, να μας κρατήσουν εκεί, εχμάλωτος. Τι είναι αυτά. Ευρωπαίους πολίτες δεν θα πρέπει εμείς να τους ε, φυγαδεύσουμε από εκεί. Το λέω σχηματικά. απαγωγή δεν είναι. Ισπανός πολίτης που τον έχουν ε, αρπάξει εκεί και κάπου τον έχουν πάει μέσα στην έρημο και δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Ισπανία. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Τι να πω. Όλα τα επιχειρήματα είναι σωστά. Απλώς θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι σωστές δράσεις. Ξέρουμε πώς γίνεται αυτό. Ε, με το Πολυσάριο μιλάμε, παίρνουν και αναπτυξιακή βοήθεια κτλ. Δεν μπορούμε εμείς να δίνουμε μια ηθαγένεια σε κάποιον που να μην αξίζει τίποτα. Είναι και θέμα εμπιστοσύνη απέναντι στι γυναίκε που είπαν συνειδητά ότι θέλουμε να γίνουμε πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χρειάζονται βοήθεια και καλά κάνουν και τη ζητάνε. Το υποστηρίζουν οι συνάδελφοι. Για φανταστείτε να μας είχαν εμά εκεί πέρα κάπου στην έρημο, εμάς τους τέσσερις και να μας είχε ξεχάσει το σύμπαν. Πραγματικά χρειαζόμαστε ε, φοδρή και στεναρή αντίδραση. Και χρησιμοποιήστε όλους τους πολιτικούς διάβλους που υπάρχουν αρκετοί δόξα τω Θεώ και να ε, απελήσουμε ότι θα τους κόψουμε και τα κονδύλια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δικοί μας ε, Ευρωπαίοι πολίτες είναι και γυναίκες, θα τους αφήσουμε εκεί μέσα στην έρημο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τέρη Καβράς. Sorry. Thank you, Chair. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το θέμα από κοντά, τις περιπτώσεις που μας αναφέρετε, αλλά μου φαίνεται εξωφρενικό αυτό που άκουσα. Όλη αυτή η αφήγηση και εξιστόρηση Συμφωνώ λοιπόν με τα εξής. Πρώτον, να διευκρινιστεί η κατάσταση. Γιατί να δούμε ποιοι είναι αρμόδιοι που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεύθυνοι, οι οικογένειες, το μέτωπο Πολυσάριο, όλοι μαζί. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεύτερον, μέχρι ποιου βαθμού έχει παρέμβει η Ισπανία. Γιατί δεν το γνωρίζω και δεν το κατάλαβα κιόλα. Ή καθόλου, ή όχι επαρκώς ακόμα που και αυτό θα ήταν σοβαρό, γιατί πρέπει να επέμβει. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, μια μικρή παρατήρηση για τις σχέσεις παιδιών με γονείς. Οι γονείς είτε είναι βιολογικοί είτε είναι άδοχοι και τα παιδιά είτε είναι ε, ανήλικα είτε ενήλικα έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τους γονείς. Και καμιά φορά αυτό το, το βλέπουμε στρεβλά. Λένε ορισμένοι ότι οι γονείς έχουν δικαιώματα επί των παιδιών τους. Όχι, τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Και αυτοί που έχουν υποχρεώσει είναι οι γονείς. Οπότε, αυτό είναι ένα θέμα απολύτως κεφαλαιόδες. Δικαιώματα έχουν ε, τα κορίτσια αυτά που είναι παιδιά, δεν ξέρω, βιολογικά υιοθετημένα ανάδοχα. Αυτά έχουν τα δικαιώματα και αυτά θα πρέπει να προστατέψουμε, γιατί οι υπόλοιποι έχουμε υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα. Δικαιώματα έχουν τα παιδιά. Κάτι που επίσης δεν κατάλαβα ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πώ θα δράσει τώρα η Κομισιόν. Δεν το κατάλαβα. Δεν λέω ότι δεν είναι σαφές. εμένα δεν μου έγινε σαφές. Τι θα έχουμε τώρα, κάποιες χειρονομίες ε, συμβολικές και ωραίες και συμπαθείς και τα λοιπά και πόσο τις αγαπάμε και πόσο ελληνική έχουμε. Αυτό θα είναι σε τέτοιο επίπεδο ή μπορούμε να ασκήσουμε πίεση γιατί πρέπει να το κάνουμε. Σε εκείνους που ήταν η ρίζα του προβλήματος, δεν ξέρω αν είναι οι ή το πολυσάριο και αυτούς που θα πρέπει να επέμβουν η Αλγερινή, η Ισπανική κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε αυτές οι γυναίκες, οι κοπέλες να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν δύο δικαιώματα. Πρώτον, να αποφανθούν οι ίδιες αν θεωρούν ότι ε, τις έχουν ε, ε, ή όχι. Εντάξει, το είπα να το επαναλάβουν. Και δεύτερον, αν ισχύσει αυτό, να έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία. Αλλά τι θα κάνουμε εμεί για να πιέσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank Ευχαριστώ, η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή τη μικρή, γιατί ήμουν αλλού. Στην αναπτυξιακή βοήθεια. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υποστηρίζουμε απολύτως τις αναφέρουσες και ε, το γεγονός αυτό στην Ισπανία και στη δική μου περιφέρεια είχαμε τέτοιες περιπτώσεις με ε, ε, νέες κοπέλες που είτε έμεναν στην Ισπανία είτε ερχόταν κάθε καλοκαίρι να πέρασουν τις διακοπές τους. Κάποια στιγμή σταμάτησε αυτό γιατί τους το απαγόρευσαν. Και μάλιστα παρά τη θέλησή τους. Και μάλιστα πρόκειται για ενήλικες. και στο όνομα μιας τοποθέτησης πολιτιστικής, πολιτισμικής, ξέρω εγώ, θρησκευτικής, καμία σχέση. Όλα αυτά με ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί βλέπω τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχω εγώ και την ενημέρωση, στο φάκελο βλέπω την Επιτροπή Γυναικών του Κοινοβουλίου που μας απάντησε και έχει προτάσεις αλλά υπάρχει και η Επιτροπή Ντρουά Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή Εξωτερικών που δεν μας απάντησαν. Και ποια είναι η πρόταση. Και ζητώ συγγνώμη που δεν άκουσα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλλον θα τα είπε. Αλλά θα ήταν σημαντικό να δούμε τι συνέχεια θα δώσουμε σε αυτές τις αναφορές και πώς θα βρούμε κάποια λύση. Και μετά, σε κάποια από τα κείμενα που διαβάσαμε, βλέπουμε το Πολυσάριο να εμφανίζεται ως συνομιλητής μας. Ξέρουμε ότι μιλάμε με το Πολυσάριο για άλλα θέματα πολιτικά αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει κανένας τρόπος εσείς ως πρόεδρος να απευθυνθείτε και στο Πολυσάριο και να εκφράσετε την ανησυχία σας. και να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Μέσω της είπα της αρμοστίας, του ΟΗΕ, δεν ξέρω, μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας, για να λυθεί αυτός ο κόμπος. Αυτές οι γυναίκες πραγματικά είναι τρομερό να κρατούνται παρά τη θέλησή τους. Και οι οικογένειες που τις έχουν ε, αναστήσει να με τις βλέπουν. Έχουν έρθει εδώ, πήγαιναν σχολείο, σπουδέ, είχαν προβλήματα υγεία, που τους βοήθησαν ε, και τις έχουν χάσει αυτές οι οικογένειες. Πραγματικά ζουν μέσα στην αγωνία και το άγχος. Ούτε να τις ζουν μπορούν, ούτε να τις επισκεφθούν, ούτε τίποτα. Υποστηρίζω αυτό που είπατε. Με ποιο τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, Πρώτον, ποιοι είναι οι συνομιλητές να μας απαντήσουν όλοι τι να κάνουμε και μετά να προχωρήσουμε, να δρομολογήσουμε κάποιες εξελίξεις. Ευχαριστώ. This is very, very difficult. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, πράγματι. Μπορούμε και πάλι να δώσουμε το λόγο στην αναφέρουσα, την κυρία Μαρία Ελίσα Παβών Μουλέρο. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο κατόπιν των σχολείων των συναδέλφων, ευχαρίστω και μετά θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή εξ ονόματος όλων των οικογενειών. Πραγματικά σας ευγνωμονούμε για το ενδιαφέρον σας, το οποίο φαίνεται, ε, θελήσατε να μάθετε και να καταλάβετε την κατάσταση. Επιτρέψτε μου να σας πω και να σας ζητήσω με όλη τη στοργή και όλη την αγάπη. Όταν ζητούμε όλες αυτές οι γυναίκες που κρατούνται και εχμάλωτες να μπορέσουν να εκφράσουν ελεύθερα την ε, βόλησή τους, να το κάνουν αυτό εκτός των καταβλισμών, μακριά από εκείνους που τους έχουν εχμαλωτήσει. Γιατί τι λέει το Πολυσάριο, ότι μέσα στους καταβλισμούς λένε ότι ελεύθερα θέλουν να παραμείνουν. Και σας λέω ρητά και κατηγορηματικά αυτό είναι ψεύδος. Δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα μέσα στους καταβλισμούς. Οπότε σας παρακαλώ, με όλη τη ιστορία και την αγάπη, όταν βλέπετε βίντεο, γιατί θα τα δείτε, με τη μαλώμα που να λέει ότι δεν με κρατούν παρά τη θέλησή μου, καταλάβετε πώς έχει η κατάσταση ε, Πώ τράβηξαν το βίντεο. Ο αδελφό της την έχει μαγνητοσκοπήσει, που είναι εκείνο που την κρατάει χμάλωτη. Κοιτάξτε, εμεί είμαστε απλοί πολίτες και εσείς ε, μας εκπροσωπείτε και είστε η φωνή μας στο Κοινοβούλιο. Σας ζητώ και σας ζητούμε τα λόγια αυτά να μετατραπούν σε έργα όλα. Και πραγματικά από κοινού να οικοδομήσουμε κάτι γιατί μπορούμε να τις βοηθήσουμε, να χτίσουμε μια γέφυρα για την ελευθερία τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολλά για όλα όσα έχετε κάνει ως τώρα. Καταρχάς ε, που φροντίσατε τα κορίτσια και μετά υποστήριξαν, υποστήριξατε τόσο πολύ τις οικογένειές τους και προσπαθήσατε με κάθε τρόπο να ε, ρίξετε φως στην υπόθεση. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να συνοψίσω. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ε, τα γυναίκες αυτές έχουν ε, δικαιώματα όπως ε, είπαν και οι συνάδελφοι νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε μια επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση Έχουμε ζητήσει και στο παρελθόν γνωμοδότηση από την Επιτροπή Γυναικών, από την Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μόνο η γυναικών απάντησε και δεν ε, μας λένε συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι λοιπόν χρήσιμο να έρθουμε πάλι σε επαφή με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Εξωτερικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγγνώμη. Ε, ε, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ένας διμερής διάλογος ε, ε, προφανώς υπάρχει διμερής διάλογος μεταξύ Ισπανίας και Αλγερία σε όλα τα επίπεδα. Να ε, το να ενισχύσουμε λοιπόν και να ενθαρρύνουμε το διάλογο αυτό είναι καθήκον τη Ισπανίας αυτή τη στιγμή. Ε, να στραφώ και προς την κυρία Μογκερίνη να προσπαθήσει να μεσολαβήσει και να ε, πιέσει για εξελίξεις στο θέμα με κάθε επαφή την οποία έχει και επίση θα ήθελα να ε, σταλεί και μία επιστολή στο Πολυσάριο δεν είναι κάτι που κάνουμε συχνά, αλλά πρέπει να ε, μάθουν ότι υπάρχει αυτή η αναφορά και ότι προσπαθούμε με κάθε δυνατό μέσο να γυρίσουν πίσω αυτά ε, τα ε, κορίτσια και να ρίξουμε φως στο τι ακριβώς του συνέβη. Νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν έχει προτείνει κανείς τίποτε καλύτερο. Αυτά τα μέσα λοιπόν μπορώ να τα προτείνω γιατί δεν έχουν ε, ακόμη ε, εξαντληθεί. Ωραία. Ούτω θα πράξουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι τις Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνατε και θα συνεχίσετε να κάνετε. Και προς όλους εσάς να ευχηθώ καλό απόγευμα. Ολοκληρώνω τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών για σήμερα.